Κυρίε Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΙΜΚΟ, αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητό κοινό, καλώς ορίσατε. Καλώς ήλθατε σε αυτό το εργαστήρι για τους νέους κανόνες για τις συμβάσεις σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Πριν κάνω τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, θα ήθελα να καλωσορίσουμε την κυρία Ηλώνα Βόλφραμ, πρόεδρο της ε, ομάδας εργασίας της Ολλανδικής Προεδρίας για το θέμα αυτό, που ε, κάθεται εξ αριστερών μου. Το εργαστήριο το οργανώνουμε για να συζητήσουμε δύο προτάσεις που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία για την επιγραμμική πώληση ψηφιακού περιεχομένου και άλλη μία για την επιγραμμική πώληση απτών αγαθών, υλικών αγαθών με στόχο να διευκρινιστούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις με τις οποίες ε, διεξάγεται το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο προτάσεις συνδέονται με την στρατηγική για την ψηφιακή αγορά το Μάιο του 2015, οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι θα παρουσιάσει προτάσεις που θα αντικαθιστούσαν την πρόταση για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο ε, ε, για τις πωλήσει. Ε, μια πρόταση πάνω στην οποία είχαμε δουλέψει πάρα πολύ, αλλά μια πρόταση η οποία δεν έτυχε επαρκούς στήριξη στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύει ακραδάντως ότι οι δύο αυτές προτάσεις ε, ανήκουν στην απόλυτη αρμοδιότητα ε, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2014 το 50% των Ευρωπαίων καταναλωτών έκαναν διαδικτυακές αγορές, ενώ το ποσοστό το 2007 ήταν 13%. Με αιτήσιο ρυθμό ανάπτυξης 22% οι διαδικτυακές πωλήσεις λιανικής αυτών υλικών αγαθών ανέρχονται σε 240 δις ευρώ το 2014 και αυτό είναι το 7% του συνόλου του ε, λιανικού εμπορίου στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι αυτό το δυναμικό ε, μπορεί να επιτευχθεί και να ενισχυθεί έροντας τους φραγμούς και τα εμπόδια, τα αριθμιστικά, τα κανονιστικά, τα διοικητικά μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό είναι και ο σκοπός της πρότασης ε, Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν να πω ότι αυτό το εργαστήριο είναι μια πρώτη εισαγωγική συζήτηση για το θέμα αυτό και από τη στιγμή που ο χρόνος μας είναι περιορισμένος θα ήθελα και οι ομιλητές να ε, μη μακρηγορήσουν πολύ για να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Και η πρώτη που θα πάρει το λόγο είναι η κυρία Ιλώνα Βόλφραμ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 μιλήσω σε αυτό το εργαστήριο για τις δύο νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα για να σας δώσω κάποιες σύντομε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει αυτό το φάκελο αυτό το Συμβούλιο. Ε, οι προτάσεις αυτές είναι σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ψηφιακή αγορά και τα θέματα που πραγματεύονται είναι θέματα που απασχολούν καθημερινά τους Ευρωπαίους πολίτες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε υψηλότερο, στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Η Ολλανδική Προεδρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στο φάκελο αυτό, τον θεωρεί ε, απόλυτη προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αυτό το φάκελο και αν επιτευχθεί η πρόοδρος επαρκής σε τεχνικό επίπεδο, στόχος μας είναι ορισμένα ζητήματα να εξεταστούν και να ρυθμιστούν οριστικά στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων του Ιουνίου. Επομένως έχουμε προγραμματίσει πολλές ε, συσκέψεις και συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας στο Συμβούλιο τους επόμενους μήνες. Έχει ξεκινήσει η δουλειά στην ε, ε, ομάδα αστικού δικαίου. Η πρώτη συνεδρία έγινε τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και η δεύτερη συνεδρία έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο και η έκβαση των δύο αυτών συνεδριάσεων ήταν εξαιρετικά επικοδομητική. Έχουμε αποκομίσει την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη θέλουν ε, σφόδρα να προχωρήσει η εξέταση του φακέλου. Ωστόσο, οφείλω να τονίσω ότι όλα τα κράτη-μέλη ε, εξετάζουν προσεκτικά την πρόταση αυτή, τις δύο αυτές προτάσεις, και σε αυτή τη φάση βρίσκονται, στη φάση της εντελεχούς εξέτασης. Παρόλο που οι απόψεις που εκφράζουν τα κράτη-μέλη είναι ακόμα προκαταρκτικές, το ότι μοιραζόμαστε πληροφορίες στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου είναι κάτι που μας επιτρέπει να έχουμε μπορέσει να εξετάσουμε σε μία πρώτη φάση τις προτάσεις. Στην πρώτη συνεδρίαση κάναμε μια γενική ανταλλαγή απόψεων για τους γενικούς ε, στόχους των δύο νομοθετικών προτάσεων. Στη συνέχεια συζητήσαμε την αξιολόγηση αντικτύπου και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη δεύτερη συνεδρίαση η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου μπήκε πλέον στην εξέταση των προτάσεων σε βάθος. Ε, ξεκινήσαμε την εξέταση κατάρθρων δίνοντας έμφαση στους λανθάνοντες, στους κύριους στόχους του κάθε άρθρου και στα αποτελέσματα που ε, θα επιφέρει η εφαρμογή του εκάστοτε, του άρθρου. Και ε, το συμπέρασμα της συζήτησης είναι ότι είναι μεγάλη πρόκληση όλα αυτά να ε, ανταποκριθούμε νομικά ε, στις ανάγκες της ζωής σήμερα και στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε σωστά αποτελέσματα που να μπορούν να εφαρμοστούν και στην πράξη. Ως προς την οδηγία και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων ε, για το ψηφιακό περιεχόμενο καλύπτεται ε, μεγάλος αριθμός θεμάτων, π.χ. εφαρμογές, ε, ε, κοινωνικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο, μεταξύ άλλων. Άλλοι τομείς όμως είναι τελείως καινοφανείς. Τα δικαιώματα του καταναλωτή καλύπτουν και την ψηφιακή σφαίρα, όμως μόνο με περιορισμένο τρόπο. Είναι απαραίτητο λοιπόν όπως και έχει γίνει και με άλλες οδηγίες, να έχουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πολλούν διασυνοριακά. Η νομοθεσία πρέπει να προβλέπει η προστασία του καταναλωτή σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη όταν προβαίνει σε ε, διασυνοριακές αγορές. Νομίζω ότι όλοι μας είχαμε ε, προσωπική εμπειρία προβλημάτων που έχουν προκύψει όταν έχουμε παραγγείλει κάτι διαδικτυακά ή ε, όταν τελικά μας παραδίδεται ένα υλικό αγαθό που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Σε τεχνικό επίπεδο είναι σημαντικό ε, οι κανόνες να είναι φιλικοί προς το χρήστη και να είναι εύκολη η απόδειξη. Φανταστείτε για παράδειγμα σε τρία χρόνια να εφεύρει κάποιος μια νέα τεχνική εφαρμογή, κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ. Θέλουμε ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ε, να του ταιριάζουν οι κανόνες που θα έχουμε αποφασίσει και που θα έχουμε νομοθετήσει. Βέβαια πάντοτε τηρώντας και σεβόμενη της ασφάλειας, της νομικής βεβαιότητας. Εάν καταφέρουμε να έχουμε σαφείς, ξεκάθαρους κανόνες που θα πετυχαίνουν ένα σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών και των συμφερόντων των επιχειρήσεων, ε, τότε θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ε, κάτι το οποίο είναι ένα στόχος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για το Συμβούλιο, πιστεύω. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, ε, πολλές είναι οι προκλήσεις κατά τη συζήτηση αυτών των προτάσεων. Και υπάρχουν και τεχνικά δυσεπίλητα ζητήματα. Όλα αυτά τα θέματα και τα νομικά και τα τεχνικά χρειάζονται προσεκτική εξέταση και η Προεδρία των Κάτω Χωρών έχει προβλέψει μεγάλο χρονικό διάστημα για την άνετη εξέταση όλων αυτών των θεμάτων και θα, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για την πρόταση. Παρ' όλα αυτά, μας ενδιαφέρει να ακούσουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προτάσεις αυτές. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου στο δίκαιο που προστατεύει τον καταναλωτή ήταν εξαιρετικά σημαντική η Επιτροπή σας έχει ε, συντάξει έκθεση για το Ευρωπαϊκό ε, κοινό δίκαιο για τις πωλήσει και αυτό ενέπνευσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη σύνταξη της συνολικής της πρότασης για το ψηφιακό ε, περιεχόμενο. Με δεδομένο λοιπόν αυτό το σημαντικό ιστορικό ε, τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή σα για τι δύο προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσδοκούμε να έχουμε επικοδομητική συνεργασία με εσά στην εξέταση αυτού του φακέλου. Σα ευχαριστώ. Ε, σα ευχαριστούμε κύριε Βαλφρόμ. Συνεχίζουμε τώρα με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Ο κύριος Ντρικ Μάιερ είναι ο επόμενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Δικαιωμάτων του Καταναλωτού. Παρακαλώ, κύριε Μάιερ. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας. Παρακαλώ, μην ξεπεράσετε το τέταρτο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Σε ό,τι αφορά τις δύο προτάσεις θα ήθελα να πω προκαταρκτικά ότι είναι οι πρώτες προτάσεις της ε, ε, στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε γιατί ε, εξηγεί το πολιτικό σκεπτικό που στηρίζει αυτές τις προτάσεις. Για τη στρατηγική για την νέα ψηφιακή αγορά έχει στόχο την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και για τους καταναλωτές εξασφαλίζοντας μία απρόσκοπτα λειτουργούσα ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτή τη, φορά έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και οι οικονομίες ε, υφίστανται μια διαδικασία ψηφιοποίησης ε, διεξοδική, αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης μας διαφέρουν με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αν δούμε τις, ε, τους ρυθμούς ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου στην στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη-μέλη εσωτερικά είναι συγκρίσιμες. Αλλά οι διαφορές οφείλονται στους διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του διασυνοριακού εμπορίου. Εκεί, ε, στα κράτη-μέλη, έχουμε εθνικά τριπλάσιες ε, ε, αγορές σε σχέση με τις διασυνοριακές. Το ίδιο και τις επιχειρήσεις. Το διασυνοριακό εμπόριο λοιπόν δεν είναι κάτι που ενθαρρύνεται μέχρι στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και το εθνικό εμπόριο και των επιχειρήσεων ε, και των καταναλωτικών αγαθών είναι τριπλάσιο σχέση με το ηλεκτρονικό. Ε, και αυτό ε, περιγράφει και τα, περι... τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Για να δούμε τι γίνεται με την πρώτη πρόταση ψηφιακού περιεχομένου. Έχουμε μια κατάσταση όπου σε λίγε χώρε. μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι ε, κάτω χώρε και την Ελλάδα έχουμε νομοθετικέ προτάσει σχετικέ και έχουμε ειδικού κανόνε για το ψηφιακό περιεχόμενο. Όλες οι υπόλοιπες χώρες μέλη εφαρμόζουν το γενικό ενοχικό δίκαιο και έτσι χαρακτηρίζουν διαφορετικά α, διαφο τα, τις συμβάσεις. Άλλες χαρακτηρίζουν συμβάσεις αγαθών, άλλες συμβάσεις υπηρεσιών, άλλες συμβάσεις αμίσθωσης. Και όλα εξαρτώνται από το ιδιαίτερο περιεχόμενο. Αυτό έχει ένα, δημιουργεί ένα πρόβλημα ε, ετερογένειας, ανομοιομορφίας και περιπλοκότητας. Επίσης ε, και τα δίκα μέσα είναι διαφορετικά και τα μέτρα αποκατάσταση είναι διαφορετικά μεταξύ των κρατών μελών. Άλλα είναι υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά. Φανταστείτε να είστε επιχείρηση, ε, δημιουργείται όχι μόνο, αντιμετωπίζετε όχι μόνο μια περίπλοκη κατάσταση και ανομοιόμορφη, αλλά και διαφορετικού κανόνε. Όπως είπα, μερικέ χώρες ήδη έχουν ξεκινήσει την νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Και εδώ υπάρχει μια όλο και αυξανόμενη τάση μεγαλύτερης ρυθμίση, Γι' αυτό και πολλέ οργανώσεις ήρθαν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησαν να αναλάβουμε δράση πριν δημιουργηθεί μια κατάσταση με ένα τοπίο που θα χαρακτηρίζεται από 28 διαφορετικά νομοθετήματα διαφορετικών ε, πολιτικών κατευθύνσεων. Οπότε ε, μέχρι στιγμή οι νομοθεσίε είναι διαφορετικέ, το περιεχόμενο είναι διαφορετικό, το πεδίο εφαρμογή είναι διαφορετικό, αλλά έχουν ένα κοινό σημείο. Είναι όλα τα μέτρα υποχρεωτικά. Οπότε, αν είστε μια επιχείρηση που θέλει να θέσει σε εμπορία ψηφιακό περιεχόμενο σε άλλε χώρε, θα πρέπει να εφαρμόσετε διαφορετικού υποχρεωτικού κανόνε, αυτού που ισχύουν σε κάθε χώρα. Και αυτό φυσικά είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. Τώρα, ερχόμαστε στις πωλήσει, επιγραμμικές πωλήσει ε, αγαθών, υλικών αγαθών. Δεύτερη πρόταση, διαφορετική κατάσταση και διαφορετικό το σημείο αφετηρίας, γιατί εδώ έχουμε εναρμόνιση, η οδηγία του 1999 για την ε, πώληση καταναλωτικών αγαθών. Αυτή η οδηγία όμως προβλέπει μια ελάχιστη εναρμόνιση, δηλαδή τα κράτη-μέλη δίνονται να την υπερβούν και το έχουν κάνει σε διαφορετικούς βαθμούς και σε διαφορετικά σημεία. Οπότε αντιμετωπίζουμε την κατάσταση που παρά την εναρμόνιση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επιχειρήσεις αν θέλουν να στοχεύσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες σε συγκεκριμένους καταναλωτές συγκεκριμένες χώρες θα πρέπει πρώτα να εξακριβώσουν τι εθνικοί κανόνες ισχύουν, να τους συγκρίνουμε τη δική τους εθνική νομοθεσία και αν ε, ισχύει στην άλλη χώρα υψηλότερη προστασία για τους καταναλωτές, θα πρέπει να προσαρμόσει τις συμβάσεις τους και ενδεχομένω και τις τιμές των προϊόντων τους. Και αυτό είναι κάτι δαπανηρό. Και αυτό το υπερβολικό κόστος θέλουμε να το αποφύγουμε για τις επιχειρήσεις. Ποια είναι λοιπόν η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Καταρχάς διδαχθήκαμε από τα απαθήματα του παρελθόντος. Δεν ακολουθούμε πια την πορεία, την άγουσα της προαιρετικής εναρμόνισης. Έχουμε ένα περιεκτικό πλέγμα νομοθετικών διατάξεων και ακολουθούμε συγκεκριμένη ε, στοχευμένη ρυθμίση που στηρίζεται στην επίλυση των προβλημάτων. Και το βλέπετε και στις δύο νομοθετικές προτάσεις που απαρτίζονται από 20 άρθρα περίπου καθεμία. Αντιμετωπίσουμε μόνο εκείνα τα θέματα όπου εντοπίσαμε διαφορές ε, στις υποχρεωτικές διατάξεις του ενοχικού δικαίου. Και αυτές οι διαφορές κοστίζουν. Μόνο αυτά τα ζητήματα αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε και όχι άλλα. Γι' αυτό και έχουμε στοχευμένη ε, πλήρη εναρμόνιση για τα θέματα όμως μόνο αυτά. Να πω δύο λόγια και για τις δύο προτάσεις ε, λακωνικά γιατί θα μπούμε σε λεπτομέρειες αργότερα στη συζήτηση, θα ήθελα να υπογραμμίσω μια πολύ σημαντική ε, τάση που διαπιστώνουμε στην πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και ε, η εκπρόσωπος της ε, Ολλανδικής Προεδρίας, η κυρία Βόλφραμ, το ανέφερε. Θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι από τεχνολογική άποψη και να έχουμε μια διαχρονική λύση που να αντέξει στις μελλοντικέ εξέλιξεις. Θέλουμε να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου οι διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με την κατηγορία του ψηφιακού περιεχομένου να έχει διαφορετικές λύσεις. Και θέλουμε να το αποφύγουμε γιατί εξαιτίας της διαφοράς των κανόνων δημιουργούνται ε, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα για ορισμένους κλάδους συγκεκριμένου τομέα. Θέλουμε επίσης να αποφύγουμε τακτικές παράκαμψης αυτών των προτύπων ή των προδιαγραφών κατά το σχεδιασμό του προϊόντος ή της επιλογής συγκεκριμένου διάβλου διανομής προκειμένου να παρακαμφθεί η νομοθεσία. Υιοθετούμε λοιπόν μια προσέγγιση όπου είναι, που είναι περιεκτική και καλύπτει το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου. Και κάτι άλλο που εμπίπτει στην προσέγγιση μας που είναι ουδέτερη από τεχνολογική άποψη και διαχρονική, αντέχει μελλοντικέ μελλοντικές εξελίξεις, είναι το ότι περιλαμβάνουμε και ψηφιακό περιεχόμενο που, που παρέχεται έναντι των δεδομένων. Γιατί τα δεδομένα είναι το νόμισμα του σήμερα και σίγουρα και του αύριο. Γιατί λοιπόν οι καταναλωτές να έχουν λιγότερα δικαιώματα ή να στερούνται των δικαιωμάτων τους μόνο και μόνο επειδή πληρώνουμε τα δεδομένα τους, γιατί και τα δεδομένα στοιχίζουν. Και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αφύπνιση και συνειδητοποίηση των καταναλωτών ότι τα δεδομένα τους ε, έχουν ένα τίμημα και τα παρακολουθούν οι πάροχοι, οι προμηθευτές και αποτελούν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Τα data, τα στοιχεία, τα δεδομένα. Γι' αυτό και περιλαμβάνουμε όλο το συναφές ψηφιακό περιεχόμενο, γιατί θέλουμε οι καταναλωτές να έχουν συγκεκριμένα και σαφή δικαιώματα. Ε, επίσης, ε, σαφή ορισμό της ε, συμμόρφωσης θέλουμε. Να είναι σαφές πότε κάτι πάει στραβά. Και φυσικά να λάβουμε υπόψη τα σύγχρονα δικαιώματα που προκύπτουν. Και πιστεύουμε ότι με την πρόταση αυτή πραγματικά επιτύχαμε σαφή και αποτελεσματικά δικαιώματα για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα ένα ε, περιβάλλον φιλικό προς επιχειρήσεις με σαφές νομικό πλαίσιο που να μπορούν οι επιχειρήσεις να πολλούν τα προϊόντα τους σε διάφορες χώρες. Τώρα για τη δεύτερη πρόταση. Δύο στοιχεία, δύο σχόλια. Όπως είπα, ε, θέλουμε μια οδηγία ελάχιστη εναρμόνισης να τη μετατρέψουμε σε μια οδηγία πλήρους στοχευμένης όμως εναρμόνισης. Και το θέμα είναι πού θα βάλουμε τον πύχη της ε, προστασίας του καταναλωτή. Ε, με την πρότασή μας ε, έχουμε μια σαφή ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή σε 365 από, τους 500, από τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές προστατεύονται περισσότερο. Δηλαδή σαφής εντυπωσιακή αύξηση της προστασίας του καταναλωτή σε 17 χώρες. Σε 11 άλλες χώρες, σε 11 υπόλοιπες, ε, προστασία του καταναλωτή θα μειωθεί λίγο για μία από, ε, από τις χώρες αυτές και ε, για 9 σε 2%. Μόνο σε αυτές τις χώρες, αλλά για συγκεκριμένα σημεία 1 και 2 μειώνεται η προστασία, ενώ για τα υπόλοιπα σημεία αυξάνεται η προστασία. Πάντως συνολικά, ακόμη και σε αυτές τις 11 χώρες, το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή είναι συγκρίσιμο, αν όχι και υψηλότερο από το ισχύον. Τώρα, μπείτε στη θέση μιας μικρομεσαίας επιχειρήσης. Ποια θα ήταν η εναλλακτική λύση? Να πάρουμε όλες τις ε, ε, διατάξεις της προστασίας του καταναλωτή και να τις συμπεριλάβουμε σε μια νέα οδηγία. Εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας ε, του καταναλωτή σε όλες τις χώρες. Δεν το κάναμε όμως, γιατί βάλτε, μπείτε στη θέση μιας μικρομεσαίας επιχειρήσης που υποτίθεται θα πρέπει να ενθαρρύνεται για να εξαγάγει με αυτή τη βάση. Είναι δυνατό να το κάνει? με τόσο υψηλά, απόλυτα υψηλά επίπεδα προστασία. Όχι. Γι' αυτό και θετήσαμε τη δεύτερη προσέγγιση. Επίσης κάτι άλλο που συζητήθηκε εκτενώς σε πολιτικό επίπεδο. Διαφορε... Διαφορές μεταξύ επιγραμμικών ε, και offline πωλήσεων γιατί περιοριστήκαμε στις επιγραμμικές και στις εξαποστάσεις πωλήσει. Γιατί, για πολλούς και διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη αγνάγνωση του ε, Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου Πολίσεων ε, πρότεινε επαναπροσανατολισμό της, πρόσθε... της πρότασης στις επιγραμμικές και μονοπωλήσεις. Και το δεχτήκαμε αυτό γιατί οι επιγραμμικές πωλήσει προϊόντων, αγαθών, ε, αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Αυτό τι είναι η μερίδα του Λέοντος, οι επιγραμμικές πωλήσει αγαθών. Γι' αυτό και περιοριστήκαμε σε αυτές και γι' αυτό θα ήταν δυνατό να, τα μέτρα να αποκλείουν αυτές τις επιγραμμικές πωλήσει. Αυτό που δεν καλύπτεται είναι η, η πρόσωπο με πρόσωπο πωλήσει. Μας ρώτησε γιατί δεν τις περιλάβατε. Είπαμε ναι, το γνωρίζουμε, ότι η μελλοντική τάση θα είναι η διανομή μέσω ενός ε, διάβλου. Και είπαμε στην ανακοίνωση με σαφήνεια ότι θέλουμε ένα συναπές πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις πωλήσει. Αλλά από τη στιγμή που θέλουμε καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Και ακόμη δεν έχουμε ε, τα δεδομένα για τις ε, πωλήσει offline. Έχουμε τα στοιχεία για τις επιγραμμικές πωλήσει. Θα συνεχίσουμε ε, και για τις face-to-face sales, για τις πωλήσει ε, πρόσωπο με πρόσωπο και θα φροντίσουμε μετά τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων να καταλήξουμε σε ένα συνεπές νομικό πλαίσιο. Και έρχομαι στο συμπέρασμα, στο διατάφτα. Κυρίες και κύριοι, αυτό που πιστεύουμε ότι έχουμε με, με την ε, επιθυμητή έγκριση αυτών των προτάσεων θα είναι μια κατάσταση επωφελή και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Θα έχουμε ένα νέο πλέγμα κανόνων σε ολόκληρη την ε, ψηφιακή αγορά, την ενιαία ψηφιακή αγορά, κάτι που θα καταστήσει πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις, γιατί αυξάνει το πεδίο δραστηριότητά του. Επίση, οι καταναλωτέ ε, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αγορά, γιατί με υψηλό επίπεδο προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υψηλότερο από το ισχύον, θα απολαύσουν περισσότερα οικονομικά πλανεκτήματα, πιο ανταγωνιστικών τιμών και μεγαλύτερης επιλογής προϊόντων. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, δόκτωρα Στάντεν Μάιερ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Χιου Μπίλ από το Πανεπιστήμιο Warwick. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω για το ζήτημα αυτό. Ασχολούμαι με το Ευρωπαϊκό Ενοχικό Δίκαιο από το 1987. Πρόσφατα συμμετείχα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη ε, της μελέτης σκοπιμότητας για κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο επί των πολίσεων. Σήμερα όμως μιλούμε για κάτι το τελείως διαφορετικό. Μιλούμε για δύο οδηγίες οι οποίες θα εφαρμοστούν μόνο σε συμβάσεις από τις επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές, B2C και καλύπτουν τους πιο σημαντικούς μόνο τομείς της αγοράς. Είναι οδηγίες, δεν είναι κανονισμοί και θα ισχύσουν και σε διασυνοριακές συναλλαγές και σε εγχώριες συναλλαγές. Και πρόκειται για οδηγίες πλήρους εναρμόνισης και όχι ένα προαιρετικό εργαλείο. Ε, γύρουν πολύ σημαντικά νομικά ζητήματα για το ευρωπαϊκό δίκαιο πόσο πολύ προχωρούμε σε σχέση με την οδηγία του 99 και γύρουν και ζητήματα έναντι σε σχέση με την νομοθεσία των ε, κρατών μελών. Και μου ζητήθηκε να μελετήσω το τι αντίκτυπο θα έχουν στην νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το 2015 υιοθετήσαμε ε, το νόμο για την προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, θέλουμε να βελτιώσουμε την προστασία του καταναλωτή και από την άλλη θέλουμε να ενθαρρύνουμε το διασυνοριακό εμπόριο στην Ευρώπη. Ως προς τη βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο είναι πολύ σημαντική γιατί πολλά κράτη-μέλη, όπως ήδη έχει αναφερθεί, έχουν, ε, δεν έχουν νομοθεσία συγκεκριμένη. Και έτσι με την οδηγία στα κράτη-μέλη ε, θα υπάρχει πρόσβαση σε νομική προστασία για το ψηφιακό περιεχόμενο ε, και θα είναι κατάλληλη η νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Και θα υπάρξει και αυξημένη προστασία του καταλωτή, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ανέφερε και ο Δ. Στάουντεν Μάιερ, η οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο δεν θα καλύψει μόνο τα προϊόντα όπως είναι ένα DVD, αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες και υπάρχει ειδική νομοθεσία στην οδηγία διάταξη για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Ενώ ε, ο νόμος για την προστασία των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζεται μόνο στις γενικές διατάξεις για τις πωλήσει και δεν είναι καθόλου συγκεκριμένο. Και αυτό συμβαίνει και στα άλλα κράτη-μέλη. Ε, ως προς την καταγγελία μιας σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τώρα η καταγγελία αυτή πρέπει να είναι Ε, μπορεί να γίνει γραπτός, ενώ σε ορισμένα κρατημέλη πρέπει αυτό να το ε, πει το δικαστήριο. Κάτι το οποίο είναι άχρηστο για τους καταναλωτές. Κανείς δεν θέλει, ή πολύ λίγοι θέλουν να περιμένουν να αποφαθεί το δικαστήριο. Και ε, είναι και χρονοβόρο γιατί πολύ συχνά το δικαστήριο που φαίνεται ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση άρα καταγγέλλεται η σύμβαση αλλά αυτό γίνεται μέσα σε δύο μήνες, ε, δύο μήνες μετά την έκδοση της απόφασης είναι πάρα πολύ χρόνος για τον καταναλωτή. Ζητώ ε, στο σημείωμα περισσότερες εξηγήσεις για το τι είναι η αποτελεσματική θεραπεία αν θέλετε, πώς μπορεί ε, όταν παραβαίνει ο εμπορευόμενος τους όρους της σύμβασης να αποκαταστήσει τη ζημία. Φαντάζομαι ότι υπάρχει οικονομική κύρωση όταν δεν παρέχονται τα υλικά, πώς μπορεί να επανορθώσει δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατάλληλο να έχουμε οικονομικές κυρώσεις σε εμπορευόμενους οι οποίοι έχουν κατά περίπτωση παραβεί τη σύμβαση, ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Αυτό θα το εξετάσει η Επιτροπή. Επομένως, είναι ανωδική η πορεία, υπάρχουν θετικά στοιχεία στις οδηγίες και υπ' αυτή την έννοια καλωσορίζω την ύπαρξή τους. Όμως, από τη στιγμή που μιλούμε για πλήρη εναρμόνιση, αναπόφευκτα ε, θα υπάρξει απώλεια ε, προστασίας καταναλωτή στα κράτη-μέλη που έχουν ήδη υιοθετήσει ε, υψηλότερα επίπεδα προστασίας των καταναλωτών έτσι όπως προβλέπεται στην οδηγία 99, το 99. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο καταναλωτής έχει άμεσο δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, να τη λήξει και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων του. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσει ιεραρχικά ε, τα ένδικα μέσα για να έχει επανόρθωση μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση όπως θέλει και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του. Άμεσα. Και θεωρούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δουλειά μας έχει δείξει ότι οι καταναλωτές αξιολογούν αυτό το δικαίωμα ως εξαιρετικά σημαντικό και έτσι έχουν εμπιστοσύνη να δοκιμάσουν νέα προϊόντα και νέες εταιρείες, νέους εμπορευόμενους που δεν είχαν δοκιμάσει πριν. Αυτό θα το χάσουμε εάν αγκρεθούν ε, οι οδηγίες έτσι όπως έχουν. Μία άλλη απώλεια εάν ερμηνεύω σωστά την οδηγία και πιστεύω ότι την ερμηνεύω σωστά, είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επανόρθωση στην περίπτωση κατά την οποία ο εμπορευόμενος δεν συμμορφούται, αλλά η απουσία συμμόρφωσης εμφανίστηκε δύο χρόνια μετά. Έχουμε πάρα πολλά προϊόντα, αυτοκίνητα, φάρμακα, όπου ε, μπορεί να περάσουν περισσότερα από δύο χρόνια πριν φανεί ξεκάθαρα ότι το εκάστοτε προϊόν δεν συμμορφούνται με τις προϋποθέσεις. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε έξι χρόνια και είναι επαρκής αυτή η χρονική διάρκεια. Τα δύο χρόνια σαν περίοδος δεν είναι επαρκής. Να, ε, μπορεί κανείς δηλαδή να ζητήσει επανόρθωση μόνο εάν το πρόβλημα εμφανιστεί στα πρώτα δύο χρόνια. Εμείς έχουμε έξι χρόνια. Από εκεί και πέρα σε πολλά κράτη-μέλη, όπως είπε και ο κύριος Μάιερ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που να διέπει το ψηφιακό περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά, όλα τα κράτη-μέλη έχουν μια κάποια νομοθεσία σχετική. Είναι αδιανόητο ένας καταναλωτής που έχει λάβει κάτι εντελώ ελαττωματικό να τον απομακρύνουμε από τη δικαστική οδό χωρίς να υπάρχει καμία επανόρθωση τα δικαστηρία θα εφαρμόσουν κατά αναλογία το δίκαιο επί των πωλήσεων αγαθών, συμβατικών πωλήσεων, όχι ψηφιακών. Και εδώ υπάρχει ανησυχία γιατί η διάταξη που ασχολείται με το ότι το ψηφιακό περιεχόμενο δεν συμμορφούνται με τις προϋποθέσεις είναι μια αδύναμη διάταξη και θα οδηγήσει σε απώλεια προστασίας του καταναλωτή σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αν δείτε τη διάταξη για την πώληση των αγαθών και υλικών ε, ε, διαδικτυακά πρέπει τα αγαθά να ταιριάζουν με τη συνήθι τους χρήση. Όμως στην οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο προϋπόθεση, η προϋπόθεση είναι πολύ πιο αποδυναμωμένη και λέει παραθέτω. Στο βαθμό που η σύμβαση δεν ορίζει ξεκάθαρα όπου δει ε, τις προ, τα προαπαιτούμενα για το ψηφιακό περιεχόμενο, ε τότε το ψηφιακό περιεχόμενο ταιριάζει για οποιαδήποτε χρήση. Δηλαδή, ο εμπορευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει λεπτομερείς όρους της σύμβασης για να συγγράψει το δικό του ορισμό για το τι είναι αποδεκτό ως υλικό και ως ε, αγαθό. Υπό τον όρο μόνο να είναι σαφή αυτά που λέει. Νομίζω ότι ο κίνδυνος για τον καταναλωτή είναι σαφέστατος, γιατί ο μέσος καταναλωτής δεν θα διαβάσει τις λεπτομέρειες, τα ψηλά γράμματα της σύμβασης πριν συμφωνήσει με αυτή. Θεωρώ δηλαδή ότι αποδυναμώνεται η προστασία του καταναλωτή και αυτό δεν χρειάζεται. Οι εμπορευόμενοι παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο σε ε, ε, απτά μέσα όπως είναι το DVD, και σε πολλά κράτη-μέλη αυτό θεωρείται παραοχή αγαθών, υλικών και υπόκειται στην ίδια νομοθεσία. Και δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αυτό, εξ όσων γνωρίζω. Εάν όμως ο εμπορευόμενος έχει την ελευθερία να αποσαφηνίσει και να διευκρινίσει τι κάνει ένα αγαθό και τι δεν κάνει, το ίδιο μπορεί να κάνει και με το ψηφιακό περιεχόμενο. Ε, μία άλλη μείωση της καταναλωτικής προστασίας που με ανησυχεί και την απαντώ στη σχετική οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο έχει να κάνει με την αποζημίωση. Και αν κατάλαβα καλά το σχέδιο οδηγίας και πρέπει να ομολογήσω με πάσα σεβασμό στον κύριο Στάουντεν Μάιερ ότι κάθε φορά που τη διαβάζω μπερδεύομαι περισσότερο σε αυτή την παράγραφο ο εμπορευόμενος θα έχει ευθύνη μόνο εάν πλήξει το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή. Όμως, όταν το ψηφιακό περιεχόμενο δεν είναι συμβατό, μπορεί να δημιουργηθούν και άλλες απώλειες. Μπορεί να τραυματιστεί σωματικά, να έχει οικονομικές απώλειες, να υπάρξει βλάβη σε τρίτους. Δεν χρειάζεται ε, δηλαδή να θεωρηθεί ο εμπορευόμενος ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις όταν το υλικό του, το αγαθό του μόνο χαλάσει π.χ. το DVD του καταναλωτή. Μπορεί να συμβούν και άλλα πράγματα μέσω του αγαθού αυτού και θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα επανόρθωσης και αποζημίωσης. Από εκεί και πέρα. Έχουμε άδεια τελικού χρήστη που μπορεί να δώσει ο εμπορευόμενος ή τρίτο μέρος. Και θεωρώ ότι ο εμπορευόμενος θα πρέπει να πει ποια δικαιώματα θα έχει ο καταναλωτής πριν πουλήσει το προϊόν. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής θα έχει δικαίωμα σε ελεύθερες δωρεάν ενημερώσεις. Θα μπορεί να έχει νέο αντίγραφο του προϊόντος εάν κάτι συμβεί με το παλιό. Μπορεί να το επαναπολύσει ο ίδιος σε άλλους. Θα πρέπει να τα ξέρει ο καταναλωτής αυτά πριν τα αγοράζει το ψηφιακό περιεχόμενο. Εάν η πληροφορία δεν δίνεται αυτή, τότε ο βάση της οδηγίας ο καταλωτής δεν έχει δικαίωμα για επανόρθωση, για αποζημίωση. Ως προς την προστασία του καταλωτή, έχω την εντύπωση ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα αυτό. Είναι μια καλή αρχή, σχετικά ξεκάθαρη, και θα μπορούσαν να λυθούν τα προβλήματα που σας αναφέρω. Ωστόσο, πιστεύω ότι οφείλουμε να αναρωτηθούμε. Είναι αυτές οι οδηγίες ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουμε το δεύτερο στόχο που είναι η ενθάρρυνση του διασυνοριακού εμπορίου είναι στοχευμένες, αλλά η στόχευσή τους είναι εξαιρετικά στενή. Δεν νομίζω ότι καλύπτουν όλα αυτά που ανησυχούν και απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες διστάζουν να μπουν στην αρένα του διασυνοριακού εμπορίου. Ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φοβούνται το άγνωστο και αν είναι πιο ευρείες οι οδηγίες θα καλύπτουν περισσότερα παιδεία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Α, λύση και απάντηση δεν είναι μόνο το να πουλάμε στους καταναλωτές. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, B2B. Ε, μόνο έτσι θα ενισχυθεί το διασυναριακό εμπόριο και θα πρέπει να γίνει δουλειά και σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ πολύ. You, Ευχαριστούμε καθηγητά Μπιλ για τα σχόλιά σας. Μπορούμε τώρα να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί δεν είμαστε εδώ μόνο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και παρακαλώ όποιος ε, θέλει το λόγο ας ε, ε, συστήνεται κιόλα. Η κυρία Ρέντα πρώτα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν πρέπει και εμείς να συστηθούμε, μάλλον όχι. Αναρωτιόμουν, θα έλεγα ναι, λέει ο πρόεδρος. Ωραία. Γιούλια Ρέντα ονομάζομαι, μέλος των, της ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος του Γερμανικού Κόμμα κόμματος των πειρατών. Ε, αναρωτιόμουν όταν μιλούσε ο, κύριο, ο καθηγητής Μπιλ για το εύρος της πλήρους εναρμόνισης ε, σε σχέση με τις ζημίες. Η πλήρης εναρμόνιση σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι είναι αδύνατον για το κράτος μέλος να ε, δώσει οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα ε, επανόρθωσης που δεν σχετίζεται με, ε, με το ψηφιακό περιβάλλον. Και το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το πεδίο εφαρμογή του ορισμού. Τι θεωρείται ψηφιακό περιεχόμενο γιατί από τη μία έχουμε την πρόταση η οποία είναι ουδέτερη ως προς την τεχνολογία, αλλά κάνει παρόλα αυτά ένα διαχωρισμό μεταξύ από τη μια του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται ψηφιακά και του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται σε ένα απτό αντικείμενο, σε μια συσκευή. Οπότε αν δούμε και το ίντερνετ των το διαδίκτυο των πραγμάτων, το οποίο εξαιρείται, δεν υπάρχει ένα σαφές όριο μεταξύ του ψηφιακού περιεχομένου σε ένα απτό, σε μια συσκευή και ένα ψηφιακό περιεχόμενο που μπορεί ίσως να το συμπεριλαμβάνει. Δεν ε, επικαλύπτει το ένα το άλλο σε ό,τι αφορά τα, ε, τα προϊόντα τα οποία έχουν ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο, οπότε παρακαλώ ο καθηγητής Μπιλ να απαντήσει. Α, συγγνώμη, ο κύριος Μάιερ πρώτα. Ευχαρίστω να δώσω στο Χιού το, το λόγο πρώτα, αλλά εντάξει πρώτα, ας μιλήσω εγώ. Καταρχάς για το εύρος της πλήρους εναρμόνισης των ε, ζημιών. Ε, ναι, είναι οδηγία πλήρου εναρμόνιση αυτή, στοχευμένη όμω πλήρη εναρμόνιση, γιατί οι ζημίες είναι ιδιαίτερο στοχευμένη. Αρχικά, μελετήσαμε τη δυνατότητα ευρεία εναρμόνιση. Το συζητήσαμε με εμπλεκόμενου φορεί, το συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη. Και οι εμπλεκόμενοι φορεί, οι ενδιαφερόμενοι φορεί μα είπαν ότι διαφορετικέ νομοθεσίε δεν είναι το πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη μα είπαν δεν είναι απαραίτητο, οπότε δεν κάναμε πλήρη εναρμόνιση για αυτό. Έτσι όπω έχει τώρα η πρόταση, Μιλούμε για ένα αρκετά περιορισμένο σημείο και ρυθμίζεται σε αυτή την πρόταση μόνο στο βαθμό που εφαρμόζεται η ε, εφαρμόζονται οι επιπτώσεις μιας πλήρους εναρμόνισης. Οι οικονομικές ζημίες είναι αυτές που ρυθμίζονται για το hardware και το λογισμικό του καταναλωτή. Αυτό που δεν ρυθμίζεται είναι ηθικές ζημίες. Για παράδειγμα, ε, η φωτογραφία σας ε, που έχετε στο υπολογιστικό νέφος, στο cloud, είναι προσβάσιμες από όλο τον πλανήτη γιατί ο πάροχος του υπολογιστικού νέφους δεν, δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας που είχε υποσχεθεί. Αυτό που δεν ρυθμίζεται είναι έμεσες ζημίες. Ε, πήρατε κάτι, θέλετε να βγάλετε κάποιο κέρδος και το όφελος αυτό δεν ρυθμίζεται όλα αυτά τα είδη λοιπόν ζημιών δεν ρυθμίζονται και αυτό σημαίνει ότι επαφείται στο κράτος μέλος και στην εθνική νομοθεσία να τα ρυθμίσει. Το ίδιο ισχύει και για αυτό που ρυθμίζεται για το δικαίωμα σε ό,τι αφορά τις ζημίες. Έχουμε την αρχή της ζημίας η οποία καλύπτεται και λέμε ποιε είναι οι ζημίες και τι σημαίνει ζημία. Αυτό σημαίνει ότι το θύμα πρέπει να μπει σε μια κατάσταση ε, στην οποία θα βρισκόταν αν δεν υπήρχαν οι επιπτώσεις της ζημίας. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, οι συνθήκες της ζημίας, ε, είναι στενή τη ενία ευθύνη ή όχι. Είναι, υπάρχουν κάποιες άλλες ε, λεπτομέρειες, ε, αμέλεια κτλ. Όλα αυτά επαφίενται στην νομοθεσία του κράτους μέλους και δεν είναι κομμάτι του κανονισμού. Γιατί προτείνουμε αυτή τη στενή ε, συσταλτική ερμηνεία. Γιατί μελετήσαμε πολλές συμβάσεις όσο προετοιμάζαμε αυτή την οδηγία και είδαμε ότι σε πολλές συμβάσεις υπάρχει κάτι που λέγεται services credits. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει ένα λατωματικό προϊόν, σε κάποιες ε, συμβάσεις ε, δεν υπάρχει δυνατότητα ε, αποζημίωσης και απλώς σας λένε ότι τις επόμενους τρεις μήνες θα πληρώνετε λιγότερα. Ένα μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το cloud computing που μελέτησε αυτές τις συμβάσεις είπε ότι ουσιαστικά σου παρέχουν την ίδια κακή υπηρεσία αλλά για λιγότερα λεφτά. Αυτό δεν θέλουμε να έχουμε. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε να υπάρξει τουλάχιστον να ρυθμίζεται το θέμα αυτό και το, το θύμα να τοποθετείτε σε μια κατάσταση ε, στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχε υπάρξει η ζημία. Το ε, επόμενο ε, σημείο για το, για το ψηφιακό περιεχόμενο στην, σε, ένα, σε μια συσκευή, απτή συσκευή. Είχαμε τρεις επιλογές όταν υποβάλαμε την λύση που τελικά επιλέξαμε. Η πρώτη ήταν να εφαρμόσουμε τους κανόνες για τα αγαθά σε όλο το ψηφιακό περιεχόμενο σε ένα απτό μέσο. Δεύτερη επιλογή ήταν να εφαρμόσουμε τους κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και η μέση λύση ήταν να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των ε, προϊόντων, των αγαθών και του ψηφιακού περιεχομένου αυτού καθ' αυτού. Σκεφτείτε τώρα εσείς ότι είστε ο καταναλωτή. Σίγουρα όλοι θα έχετε αγοράσει μια ταινία, ένα DVD ή μουσική σε ένα, με ένα, CD. Αν, είσαστε ο, ε, δικηγόρος, αν δεν είστε ο δικηγόρος που ξέρει τα πράγματα, ε, θα είχατε σκεφτεί ότι το να κάνει κανείς μια, ένα διαχωρισμό και να βάλει διαφορετικούς κανόνε κανόνες στο πλαστικό και στο περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτό το πλαστικό θα είχε νόημα. Έχετε δηλαδή δύο κανόνες και πρέπει να κάνετε ένα διαχωρισμό που είναι το πρόβλημα και μετά να εφαρμόσετε διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με το που είναι το πρόβλημα. Ε, Κανένα ε, ε, έχει έφρον άνθρωπο δεν θα μπορούσε να σα το εξηγήσει αυτό. Και έχουμε τα δύο άκρα βεβαίω. Θα μπορούσαμε να πούμε όλα τα αγαθά ή όλο το ψηφιακό περιεχόμενο να υπόκειται στου ίδιου κανόνε. Βασικά αυτό που κάναμε και στις συζητήσεις μας αυτό είπαμε, είναι ότι ρωτήσαμε πού βρίσκεται η οικονομική προτεραιότητα, ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Η, ε, τιμή του ε, πλαστικού είναι μηδαμινή. Η οικονομική αξία είναι αυτό το οποίο ε, περιλαμβάνει το, το CD. Το περιεχόμενο λοιπόν. Οπότε είπαμε θα εφαρμόσουμε του κανόνε για το ψηφιακό περιεχόμενο και ο δεύτερο λόγο γι' αυτό ήταν ότι αν το είχαμε κάνει διαφορετικά, τότε θα είχαμε ανοίξει την πόρτα για να εφαρμόσουμε, ε, για να, ε, να οργανώσει κανεί διαφορετικά λίγο την, ε, το, τους διάβλους, τις διάβλους παροχής και να μπορεί να αποφύγει τους κανόνες. Οπότε είπαμε ότι εφαρμόζονται κανόνες για το απτό μέσο. Και είναι σαφής ο διαχωρισμός, ξεκάθαρος και συμμορφώνεται και με το οικονομικό σκεπτικό πίσω από το προϊόν και είναι και κατανοητό από τον καταναλωτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μήπως ο καθηγητής Μπίλ θα ήθελε το λόγο για να σχολιάσει πριν δώσουμε το λόγο και στους άλλους συναδέλφους. Εν συντομία θα ήθελα να πω ότι με ανακούφιση άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να αποκλείσει το δικαίωμα και σε περαιτέρω αποζημιώσεις. Αυτό όμω δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του επεξηγητικού σημειώματο. αλλά αν μα διαβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ ωραία. Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο σε ένα απτό υπόθεμα, νομίζω ότι είναι πολύ λογική η προσέγγιση Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αλλά υπάρχει και διαφορετικό τρόπο για να το πετύχουμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι το ψηφιακό περιεχόμενο, όπου και αν περιλαμβάνεται, θα πρέπει να πληρεί τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης τη οδηγίες για το ψηφιακό περιεχόμενο. Οπότε και το ε, CD και το DVD που έχουν το, από το υπόθεμα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ε, και να τα μεταχειριστούμε ως αγαθά που οφείλουν να συμμορφώνονται με την οδηγία. Αυτό όμως δεν υπάρχει στην παρούσα οδηγία. Τι γίνεται με ένα μηχάνημα που έχει εσωματωμένο λογισμικό και που έχει σχεδιαστεί να μιλά σε, άλλα, ε, σε άλλες Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και το εσωματωμένο λογισμικό θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας για το ψηφιακό περιεχόμενο. Πάντως οι ιδέες της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής έχουν απόλυτη λογική. Ο κύριος Μάγερ. Βέβαια το εσωματωμένο λογισμικό είναι πολύ σημαντικό θέμα, όπως είπε και η κυρία Ρέντα, ε, για όλο και περισσότερα ε, το διαδίκτυο των πραγμάτων που αποκτά όλο και μεγαλύτερε διαστάσει. Θέλουμε μια ρεαλιστική διάκριση. Αυτό που λέμε στην οδηγία είναι ότι όταν έχουμε ενσωματωμένο λογισμικό που αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα του αγαθού και οι λειτουργίες του υπόκεινται στις γενικότερες λειτουργίες του αγαθού, ισχύουν οι ε, υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, ένα πλυντήριο ε, Φυσικά και σε ένα πλυντήριο ρούχων, όπως και σε άλλες συσκευέ, υπάρχει λογισμικό που στόχο έχει να κάνει την, το πλυντήριο να πλένει. Αν κανείς αγοράσει ένα πλυντήριο που δεν πλένει, που δεν δουλεύει, πηγαίνει στο λιανέμπορο και λέει κάντε το να ε, δουλέψει, κάντε το να πλύνει. Δεν σκέφτεστε το λογισμικό. Πάντως, εδώ έχουμε ένα σωματωμένο λογισμικό αναπόστατο στο τμήμα της οικιακής συσκευής που εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της ε, ε, συσκευής. Και για αυτό το λογισμικό ισχύουν υποχρεώσεις ε, και που ισχύουν και για το αγαθό. Σκεφτείτε τι λογισμικό έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Τέσλα. Τεράστιο. Πάντως, ε, σκοπός του είναι να στηρίξει τη λειτουργικότητα του αυτοκινήτου, που είναι να μεταφέρει από το σημείο Α στο σημείο Β. Βέβαια, στο μέλλον μπορεί αυτό να αλλάξει. Αλλά τα επόμενα 10-15 χρόνια είμαστε ασφαλείς και έχουμε ρεαλιστική διάκριση για το εσωματωμένο λογισμικό, το οποίο θα πρέπει να πληρεί και τις ίδιες υποχρεώσεις που πληρούν και τα αγαθά. Και νομίζω ότι υπάγονται όλα αυτά στην κοινή λογική. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις και σύντομες απαντήσεις. Ο κύριος Αξελφός που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το ψηφιακό περιβάλλον. Έχουμε το μεταξύ πάρα πολλές συμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την παροχή μιας υπηρεσίας και ως αντιπαροχή να λάβουν τα δεδομένα. Αν έχουμε μια τέτοια συμβατική σχέση μία διεκπαιρέωση αυτής της σύμβασης πώς γίνεται. Δηλαδή τα δεδομένα, αν κάποιος δεν τα δώσει, τι γίνεται. Έχουμε από τη μία τον, τη χρήση του αντικειμένου της σύμβασης, αλλά από την άλλη αν αυτό το αντικείμενο της σύμβασης δεν δεν είναι χρηστικό πλέον ή είναι λατωματικό και πρέπει να υπάρξει κάποια ε, διόρθωση. Ε, τι γίνεται με, τον, ε, με τα δεδομένα, γιατί ο καταναλωτής ουσιαστικά δεν μπορεί να πάρει πίσω τα δεδομένα του, Οπότε θα ήταν καλό ίσως να μας διευκρινίσετε λίγα τι γίνεται σε μια τέτοια σχέση, όπου η παροχή είναι η υπηρεσία και η αντιπαροχή είναι η χρήση δεδομένων. Ναι, και άλλο ένα ερώτημα από τον Λόρδο Oates, από τη Βολή των Λόρδων. Um, Ευχαριστώ. Μιλώ εξ ονόματός μου βέβαια και όχι εξ ονόματος κάποιου άλλου, αλλά πρέπει να πω ότι το ε, Ηνωμένο Βασίλειο ε, καλωσορίζει τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάποια θέματα ήθελα και εγώ να θίξω, κάποια τα τόνισε ήδη ο καθηγητής Μπιλ, κυρίως σε σχέση με το μίσο όπου οι προτάσεις θα αδικατόπτριζαν μία, υπον, θα διήλυζαν λίγο την, ε, την ουσία της, ε, της πρότασης. Ε, το είπε και ο καθηγητής Μπίλ για, την, για το δικαίωμα στην άμεσο τερματισμό μιας σύμβασης. Εμείς στον Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μία εξαιτή περίοδο μέσα στην οποία μπορεί κανείς να έχει αποζημίωση για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλά για δύο χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κατανοεί βεβαίως ότι για τους εθνικούς ε, βουλευτές ε, είναι δύσκολο να ε, εξηγήσουν στο εκλογικό τους κοινό μια τέτοια διαφορά. Και ένα ερώτημα έχω που σχετίζεται με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων για το ελεύθερο περιεχόμενο, το δωρεάν περιεχόμενο. Για να καταλάβουμε λιγάκι καλύτερα πώς θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι προτάσεις αυτές είναι αναλογικές και δεν ε, είναι επιζήμιες σε αυτό που μπορεί να είναι χαμηλού ε, ε, έτσι, περιθωρίου, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί αντικείμενο επιχειρησιακών μοντέλων. Ευχαριστώ. Και ένα ερώτημα από την κυρία Γκέπχαρτ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε και τη δική μας ε, επιτροπή. Εγώ βέβαια είμαι και μέλος της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, οπότε είμαι έτσι σχετικά ε, σε μια εύκολη κατάσταση εδώ. Τρία σημεία ήθελα να τονίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικά για μένα, για την συζήτηση που κάνουμε για αυτό το τομέα. Το ένα είναι ότι χρειάζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Θέλουμε οι πολίτες μας ε, να ε, θεωρούν ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το ευρωπαϊκό όρομα είναι κάτι θετικό. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα πολύ σημαντικό, ε, να θέσουμε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε και ο εκπρόσωπος της Βουλής των Λόρδων, δεν θυμάμαι το όνομά του, ζητώ συγγνώμη, γιατί μόλις είπε ότι κάποια κρατημέλη σε κάποιους τομείς έχουν πολύ υψηλότερη προστασία ε, σε σχέση με αυτή που παρέχεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πάντα δύο δυνατότητες για να το απαντήσει κανείς αυτό. Η μία είναι να πει ότι ναι θα πάρουμε το υψηλότερο ε, ε, το επίπεδο προστασίας που υπάρχει αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό περίπτωση να εφαρμοστεί ή θα πούμε ότι θα κάνουμε αυτό που ε, ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, μια στοχευμένη εναρμόνιση ή μια ελάχιστη εναρμόνιση, έτσι ώστε το δίκαιο που είναι υψηλότερο σε κάποια κρατημέρη να μπορεί να διατηρηθεί το δίκαιο που παρέχει υψηλότερη προστασία. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο μου σημείο. Οι κανόνε του Ρώμη 1, που ε, είναι πολύ σημαντικοί για του καταναλωτέ, θα πρέπει να διατηρήσουν την ισχύ του. Κάτι που δεν θα ίσχυε αν, όπω το προτείνει τώρα εδώ η Κομισιόν, έχουμε πλήρη εναρμόνιση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί και να, ε, πάμε, να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά με αυτές τις διατάξεις. Τρίτο σημείο είναι το θέμα της νομικής ασφάλειας της νομικής ασφάλειας για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους καταναλωτές. Και θα πρέπει να φροντίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν ε, διαστρεβλώσεις ε, έτσι ώστε κάτω από κάποιες συνθήκες να υπάρχει διαφορετικό δίκαιο για τα απτά αγαθά και για τα μη ε, απτά, το ψηφιακό περιεχόμενο. Θα πρέπει δηλαδή να μην μπορεί να ορίσει κανένας κάτι όπως θέλει. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά, να δούμε ποια άγουσα θα ακολουθήσουμε. Και στην έκθεση που έχει υποβληθεί από την κυρία Κάλλα και εμένα, ήδη από τι 19 ε, Ιανουαρίου και που έχει ψηφιστεί, είχαμε πει σαφώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διαγορισμός. Θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο δίκαιο, η ίδια νομοθεσία, γιατί αλλιώ τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Φανταστείτε, α πούμε, ότι κάποιο ε, παίρνει ένα, ε, ένα πλυντήριο από το κατάστημα, και ή παίρνει ένα ε, πλυντήριο από το, ε, από το ίντερνετ και ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για το μεν και διαφορετικοί για το δε. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να το κατανοήσει ένας καταναλωτής, θα τον μπερδέψει ακόμη περισσότερο και θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως οι μεγάλες επιχειρήσεις να μην έχουν τόσο πολλά προβλήματα, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται νομική ασφάλεια. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρξει διαφορετικό δίκαιο ανάλογα με το ποιο πουλάει πού. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά για μένα και νομίζω θα πρέπει να συζητηθούν λεπτομερώς. Uh, Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ σύντομε απαντήσεις, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω στο χρονοδιάγραμμα μας. Θα έχετε και αργότερα την ευκαιρία να θέσετε ερωτήσεις. Μην βιάζεστε όλοι τώρα. Ποιο θέλει πρώτα το λόγο, κύριε Στάν Μάιερ. Θα είμαι σύντομο κύριε Πρόεδρε το ερώτημα ε, του κυρίου Φως για, την, ε, ε, για τα δεδομένα ως πληρωμή. Ναι, προφανώς δεν μπορεί να δώσει κανείς πίσω τα δεδομένα, γι' αυτό η οδηγία προβλέπει ότι ο πάροχος δεν κάνει χρήση των δεδομένων πλέον. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα τα οποία έχει διαβιβάσει μετά την ε, λήξη της ε, ε, σύμβασης, αυτά μπορεί να τα, δώσει, να τα προωθήσει, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μετά την, τον τερματισμό της, της σύμβασης δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, άρα δεν μπορεί να, έχει, να κερδίσει χρήματα από αυτά. Uh, Εκτιμούμε απολύτως ότι είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς τους καταναλωτές ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι ε, θα μειωθεί το επίπεδο προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να το εξηγήσει κανείς αυτό είναι με πρακτικούς όρους. Να δει δηλαδή τα έξι, όρια, τα έξι χρόνια όριο ε, που υπάρχει στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες, ο αντίκτυπος είναι περιορισμένος. Καταλαβαίνουμε ότι μόλις 1% των καταναλωτών στη Βρετανία γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα 6 χρόνια ως όριο και σύμφωνα και με την έρευνα που κάναμε, λίγο πριν υιοθετηθεί, πριν η πρόταση, 50% ε, των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι η εγγύηση κρατάει ένα χρόνο και ίσως ε, δύο χρόνια το πολύ. Οπότε θεωρητικά ε, πιστεύουν αυτό που προτείνει η οδηγία. Γι' αυτό η οδηγία είναι και λογική. Και επίσης η, προ... πλειοψηφία θεωρεί ότι για τις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες, ε, τα λευκά είδη, τα καφέ και τα γκρι, είναι η το σωστό χρονικό όριο. Οπότε δεν θα έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Τώρα, Υπάρχει και η συμβολική αξία, ναι, το κατανοούμε, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη και ότι η οδηγία για την προσθέτωση των καταναλωτών δίνει τη δυνατότητα ε, των, ε, των δύο εβδομάδων. Για την τρίτη και την τέταρτη ε, εβδομάδα μιλούμε. Εκεί προκύπτει η διαφορά. Σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα, οι καταναλωτές σε μεγάλη πλειοψηφία πάνε πίσω μετά από λίγες μέρες τα προϊόντα τους και το πολύ μέσα σε μια εβδομάδα. Οπότε η τρίτη και η τέταρτη εβδομάδα στην πράξη δεν, ε, ε, δεν ισχύουν, δεν ε, χρησιμοποιούνται ποτέ. Και ξέρω ότι είναι πολύ, πολύ ρεαλιστές οι Βρετανοί πολίτες και αυτό θα ήταν ένας καλός ε, τρόπος για να το διαχειριστούν για το δικαίωμα επαναχώρησης. Τώρα για το ψηφιακό δεδομένο, για το ψηφιακά το ψηφιακό περιεχόμενο και τα δεδομένα. Αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε είναι η καινοτομία μέσω νέων startups, νέων επιχειρήσεων μικρών που, που είναι καινοτόμες και δημιουργούν θέσει εργασίας. Και γι' αυτό είπαμε ότι δεν, ε, δεν μιλούμε για όλα τα δεδομένα. Ε, το έχουμε περιορίσει πάρα πολύ. Μιλούμε για προσωπικά δεδομένα, ναι, και άλλα δεδομένα, αλλά όχι ε, τα μεταδεδομένα και η ηλεκτρονική διεύθυνση, το IP ε, ούτε μιλούμε για δεδομένα τα οποία θα πρέπει να συλλέξει κανείς για να εφαρμόσει το, το δίκαιο ή που πρέπει να συλλέξει για να μπορέσει να ε, παράσχει την ε, την, ε, την ε, υπηρεσία όπως ας πούμε οι χάρτες του GPS που πρέπει να ξέρουν πού είναι το σημείο που βρίσκεστε. Έτσι η πρότασή μας ως προς αυτό είναι αναλογική. Για, την, για τα κριτήρια της συμμόρφωσης. Το πρώτο κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι έχει διαφορά αν δίδεται έναντι αμοιβή ή έναντι δεδομένων. Αυτό λαμβάνεται υπόψη. Οπότε συνολικά θεωρούμε ότι είναι ισόρροπη η προσέγγιση μας. Κυρία Γκέφχαρτ η υψηλή ε, προστασία των καταναλωτών. Ναι, έχουμε την ίδια άποψη, είναι πολύ σημαντική. Είπατε κι εσείς ότι το ανώτατο ε, ε, επίπεδο προστασίας δεν θα είχε καμιά πιθανότητα εφαρμογής. Αυτό βλέπουμε κι εμείς. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι θα έχουμε έναν σωστό, ένα στόχο της πρότασης, τον οποίο μάλλον δεν θα επιτύχουμε. Δηλαδή, η, η ε, μόνο με πλήρη εναρμόνιση θα μπορέσουμε να επιτύχουμε οι επιχειρήσεις να ε, δρούν, ε, να δραστηριοποιούνται μόνο με, ένα, με μία νομοθεσία, σύμφωνα με μία νομοθεσία, γιατί αλλιώς θα ήταν δυνατό να επιτύχουμε και το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, που είπατε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Η ελάχιστη λοιπόν εναρμόνιση είναι καλή για τους καταναλωτές και ήδη έχουμε υψηλή, υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών, αλλά για τις επιχειρήσεις δεν θα είναι αρκετά επιτυχές ή όσο επιτυχές θέλουμε να είναι. Για τους κανόνες της Ρώμης 1. Μάλλον υπάρχει κάποια παραξήγηση εδώ. Οι κανόνες της Ρώμης 1 εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Θα, τις, θα τους εφαρμόσουμε, θα συνεχίσουμε να τους ε, εφαρμόζουμε. Δεν ε, αλλάζει αυτό. Άρθρο 6, παράγραφος 2 μιλάει για πλήρη εναρμόνιση και δεν, ε, δεν έχει ισχύ πλέον γιατί οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Άρα δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω αν εναρμονίσουμε σε υψηλό επίπεδο τους κανόνες. Οπότε μετά δεν ε, έχει, δεν έχει σημασία αν το 6-2 έχει ψηλότερο, παρέχει ψηλότερο επίπεδο προστασία. Το θέμα είναι να βάλουμε τον πύχη ψηλά. Και επίση, νομική ασφάλεια συμφωνούμε απολύτω και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ξεκάθαρα στην ανακοίνωση που έχει υποβάλει ότι δική μας, ο δικό μα στρατηγικό στόχο είναι να έχουμε ένα ενιαίο ε, νομικό πλαίσιο για όλα τα αγαθά. Τα, τα, τα απτά, τα offline, τα online, απλώ τα δεδομένα θα τα συμπεριλάβουμε στην όλη διαδικασία ε, νομοθεσίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά Μπίλ, παρακαλώ, χρόνο φίδου. Ο κύριος Σταν Μάιερ ε, και εγώ θα μπορούσαμε να φιλερούμε για ώρες ολόκληρες. Καλύτερα να δώσουμε το χρόνο και στους υπόλοιπους ομιλητές να λάβουν το λόγο και αν μείνει στο τέλος χρόνος ε, θα δευτερολογήσω και εγώ. Ναι, όντω. Θα έχουμε και αργότερα ευκαιρία για συζήτηση περαιτέρω. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην καθηγήτρια Βανέσα Μάρκα από το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ και στον καθηγητή Γιάν Σμιτ από το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ. Δέκα λεπτά και οι δύο μαζί όμως. Ευχαριστώ. Δέκα λεπτά μας το ότι έχουμε ο καθένας όμως. Όχι, όχι, λάθος δικό μου. Δέκα λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Βανέσα Μάκα ονομάζομαι, είμαι καθηγήτρια ιδιωτικού δικαίου στο ε, Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ και ο καθηγητής Σμιτ και εγώ Σχολιάσαμε όπως μας ζητήθηκε τις διάφορες διατάξεις των ε, δύο προτάσεων. Χωρίσαμε τη δουλειά μεταξύ μας έτσι ώστε ο καθηγητής Σμιτ να σχολιάσει για την, ε, για την πώληση την επιγραμμική των αγαθών και εγώ θα επικεντρωθώ στο, στην πρόταση για, την, ε, για το ψηφιακό περιεχόμενο. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που μας δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσουμε εδώ τις απόψεις μας. Κατανοώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα προς συζήτηση για την πρόταση και γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε μερικά σημεία και θα σας παραπέμψω στο ενημερωτικό έγγραφο που υπάρχει για τα υπόλοιπα. Τα ε, πέντε σημαντικά σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω βρίσκονται στη διαφάνεια και κάποια ήδη έχουν προκύψει και στις ε, ερωτήσεις που ετέθησαν, οπότε νομίζω ότι είναι καλή στιγμή αυτή για να διευκρινίσουμε λιγάκι κάποια σημεία. Καταρχάς να δούμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Το θέμα αυτό ε, αναφέρθηκε ήδη. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή, όπως είπε και ο καθηγητής Μπίου, να έχουμε την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο και αν μπορέσουμε τελικά να έχουμε κάτι που θα έχει και μια ε, λύση που θα δίνει μια προστασία για το μέλλον και με παροχή προστασίας του καταναλωτή, θα είναι πολύ χρήσιμη και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Τι σημαίνει όμως προστασία για το μέλλον, αν δείτε τον ορισμό του ψηφιακού περιεχομένου στο άρθρο 2.1 βλέπουμε ότι το περιεχόμενο αυτό αναφέρεται, ε, ορίζεται με τρεις πρώτους. Ο πρώτος ε, είναι αρκετά ευρύς. Λέει ότι μιλούμε για δεδομένα τα οποία παράγονται σε ψηφιακή μορφή όπως ε, βίντεο, ηχητικά εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια και άλλο λογισμικό. Μετά βλέπουμε τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δημιουργία, την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων σε ψηφιακή μορφή όπου, που νομίζω ότι εδώ είναι οι υπηρεσίε του υπολογιστικού νέφους για παράδειγμα και μετά έχουμε την υπηρεσία που επιτρέπει την ε, ανταλλαγή και την διάδραση με δεδομένα σε ψηφιακή μορφή όπως ας πούμε σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά φαίνονται αρκετά ε, ευρεία και μπορεί όντω να παρέχουν την απαραίτητη προστασία για το μέλλον, αλλά έχουμε κάποιε ανησυχίε για το πόσο, είναι αυτός, πόσο εφαρμόσιμος είναι αυτό ο κανονισμό. Αυτό ήδη φύγει από την ε, κυρία εδώ στα ε, δεξιά, δεν βλέπω το όνομά τη, αν μπορούμε να κάνουμε έναν ε, διαχωρισμό μεταξύ των φυσικών αγαθών και των ψηφιακών αγαθών, κυρίω σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο των πραγμάτων, νομίζω ότι ε, ο ορισμός της οδηγίας ε, είναι ε, λειτουργικός. Ο ορισμός λέει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο στα αγαθά με τέτοιο τρόπο που να λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του αγαθού και, τα, και οι λειτουργίες του υπόκεινται στις λειτουργίες του αγαθού. ας πούμε, ένα αυτοκίνητο Τέσλα όπως είπε και ο κύριος Στάουτμαϊερ πριν. Έχουμε το software ενσωματωμένο στο αγαθό, στο αυτοκίνητο. Μπορεί να υπάρχει ένας διαχωρισμός εκεί, θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι κάποια αγαθά έχουν μια λειτουργία που είναι πιο προφανής από τη λειτουργία του ψηφιακού περιεχομένου, αλλά εμείς δεν είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση αυτός ο διαχωρισμός ή ότι θα είναι ξεκάθαρος ακόμη και αν γίνει στους καταναλωτές. Σε ποιε περιπτώσεις δηλαδή υπάρχει ο διαχωρισμό και πού όχι. Αν δείτε το, Tesla, το αυτοκίνητο Tesla, ναι είναι ένα αυτοκίνητο και ο σκοπό είναι να μπορεί να το οδηγήσει κάποιο, αλλά έχει τόσο πολύ ενσωματωμένο software στο αυτοκίνητο που, μπορεί να οδηγηθεί, που δεν μπορεί να οδηγήσει κανείς χωρίς αυτό το software. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα όπου το software είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του προϊόντος, του αυτοκινήτου εμπροκειμένου. Και εδώ είναι καλός ο, ορισμός που υπάρχει και το διαχωρισμό που γίνεται μεταξύ των απτών αγαθών και του ψηφιακού περιεχομένου. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, όπως είπε ο καθηγητής Μπίου, καλό είναι να έχουμε όλο το ψηφιακό περιεχόμενο ε, να εμπίπτει στους κανόνες της ε, οδηγίες έτσι ώστε να υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις δυνατότητα προστασίας του καταναλωτή. Ακόμη μία λύση θα μπορούσε να ήταν να υπάρξουν συγκεκριμένοι κανόνες για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Βεβαίως αυτό θα σήμαινε περισσότερη δουλειά για τις τρέχουσες προτάσεις, για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν αυτοί οι κανόνες και η ε, Κριστιανά Φάντερ Χόρστ που θα μιλήσει αργότερα σήμερα έχει ήδη κάνει κάποιες ε, προτάσεις, οπότε σας παραπέμπω στη δική της ε, δουλειά προς το παρόν σχετικά. Άλλο ένα ερώτημα που έχω σε σχέση με τον ορισμό είναι τι σημαίνει δεδομένα που παράσχονται από τον ε, καταναλωτή. Αν δούμε την, ε, τα δεδομένα που παράσχονται από τον καταναλωτή, Αυτό θα μπορούσε να είναι τμήμα και του ψηφιακού περιεχομένου. Η οδηγία ορίζει ότι αυτό, θα, αυτό σημαίνει δεδομένα που έχουν ενεργητικά ε, παρασκευθεί από τον καταναλωτή. Κατανοώ βεβαίως από αυτό που είπε ο Στάντον Μάιερ ότι ε, έχουν υπάρξει συζητήσεις για το πώς μπορεί κανείς να, προ... να καταλήξει μια προσέγγιση ισόρροπη, αλλά αναρωτιέμαι, γιατί συμπεριλαμβάνουμε μόνο δεδομένα που παράσχονται ενεργώς από τον καταναλωτή. Μία αντιπαροχή ας πούμε δεν θα μπορούσε να υπάρχει με δεδομένα που δεν έχουν ε, παρασχεθεί ενεργώς, ας πούμε τις ε, διευθύνσεις IP ή τα μεταδεδομένα, δεδομένα δηλαδή που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει το ψηφιακό περιεχόμενο. Και τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου η αντιπαροχή υπάρχει με μεταφορά copyright, που μπορεί επίσης να, είναι το, η που μπορεί να, επίσης να ισχύει όταν φορτώνουμε φωτογραφίες στις κοινωνικές πλατφόρμες. Έχουμε βεβαίως και το άρθρο 6.2 ε, που ε, ασχολείται με τέτοιου είδους δεδομένα. Ε, τώρα, αυτά σε σχέση με τον ορισμό του ψηφιακού περιεχομένου. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν να βελτιωθούν. Μάλλον χρειάζεται απλώς λίγο χτένισμα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα άλλο θέμα είναι η αντιπαροχή που δεν έχει να κάνει με την καταβολή μιας τιμής. Το είπε και ο κύριος Φως. Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί, να συμπεριληφθεί αυτό στην πρόταση. Νομίζω ότι θα προσθέσει πολλά, θα εμπλουτίσει σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, αλλά με ποιο τρόπο θα πρέπει να το διαχειριστεί αυτό η πρόταση. Πώ διαχειρίζεται δηλαδή η πρόταση μια τέτοια σύμβαση. Ένα ερώτημα που ε, προέκυψε όταν ε, δουλεύαμε την πρόταση αυτή είναι τι περιμένει ο καταναλωτή από πλευράς προστασίας από τη μη συμμόρφωση με το ψηφιακό περιεχόμενο. Έχει υπάρξει μια, μια πρόταση ότι αν το ψηφιακό περιεχόμενο δοθεί δωρεάν, όπου τα δεδομένα θεωρούνται ως κάτι που παρέχεται δωρεάν, ε, τότε η ε, προσδοκία του καταναλωτή σε ό,τι αφορά την συμμόρφωση μπορεί να είναι πιο χαμηλή για τέτοιου είδους προϊόντα. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι αυτό είναι ο τρόπο, ο σωστό τρόπο να αξιολογήσουμε την κατάσταση, γιατί πολλοί καταναλωτέ γνωρίζουν ότι δεν δίνοντα τα δεδομένα του ε, δίνουν κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Οπότε για αυτέ τι περιπτώσει ίσω οι καταναλωτέ θα έπρεπε να λαμβάνουν την ίδια προστασία. Αν, ε, όπως θα λάμβαναν αν έδιναν κάτι επιπληρωμή. Το είπε και ο κύριο Στάδων Μάιερ αυτό, ίσω να μπορούσαμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο στη συνέχεια αυτού. Αν ε, δούμε τα δεδομένα που παράσχονται ε, ε, αντί για την καταβολή τιμής και τι γίνεται με τους κανόνες της προστασίας δεδομένων αν αποσύρονται τα δεδομένα αυτά, το έκανε ο σχόλιο και ο κύριος Βος. Η συμβατική λύση που προτείνει η οδηγία αναρωτιέμαι αν ταιριάζει σε τέτοιου είδους δικαιώματα οι συμβατικέ συνέπειε ποιε θα πρέπει να είναι. Η οδηγία φαίνεται να προτείνει ότι υπάρχει το δικαίωμα της, ε, του τερματισμού και αυτό μπορεί να λύσει τέτοια προβλήματα, τέτοιου είδου περιπτώσει. Και υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία που ε, λένε ότι οι εταιρείε δεν θα μπορούν να τα διατηρούν ή να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά, αλλά να ρωτιέμαι, αυτό είναι συμβατικό τερματισμό, γιατί η ε, σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει, να υπάρχει. Ο καταναλωτή μπορεί να συνεχίσει να έχει τον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μπορεί να θέλει να αφαιρέσει όλε τι φωτογραφίε του. Η συμβατική λύση σε αυτή, υπό αυτή την ενία, συμνάδει με τα δικαιώματα προστασία των δεδομένων του. Πολύ σύντομα για το τρίτο σημείο, γιατί ήδη συζητήθηκε, ε, αναφέρθηκε από τον ε, καθηγητή Μπίουλ για τους ε, κανόνες μη συμμόρφωσης της πρότασης που είναι πολύ χαμηλότερης, παρέχουν πολύ χαμηλότερη ποιότητα σε σχέση με τους κανόνες των πωλήσεων κυρίως λόγω και του ότι είναι πολύ τεχνικά αυτά τα προϊόντα. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε μία λύση όπου θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ε, θεσμική προστασία ε, παρά την, ε, τους συμβατικούς κανόνες που παρέχουν προστασία του, παρόχου του ψηφιακού περιεχομένου. Τέταρτο σημείο αναφέρεται στην ε, ε, πρόταση που αφορά στο ψηφιακό περιεχόμενο που ε, μιλά για την αντιστροφή του βάρους απόδειξης και που θα πρέπει να είναι δυνατό για τους καταναλωτές να θεωρούν υπεύθυνο τον πάροχο για απεριόριστο χρόνο. Αν δούμε το κείμενο της οδηγίας βεβαίως δεν πρόκειται για απεριόριστο χρόνο γιατί υπάρχουν και εθνικοί κανόνες που ορίζουν την, τους την περίοδο αυτή ευθύνης. Και το ερώτημα είναι γιατί η οδηγία δεν, συνα... δεν υποβάλλει τους δικούς της κανόνες σχετικά. Στην πράξη φαίνεται μάλλον απίθανο οι καταναλωτές να θέλουν να θεωρήσουν υπεύθυνο έναν πάροχο για πάρα πολύ καιρό, χωρίς όριο, ε, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα που ο καταναλωτή δεν, δεν θα ενδιαφέρεται να έχει ε, να, πάρει κάποια αποζημίωση μετά από 5-6 χρόνια. Ούτως ή άλλως ε, υπάρχει ένα τέτοιο όριο τους ή ε, όλος υπάρχει ένα τέτοιο όριο που προβλέπεται. Η υπάρχουν υπαρχει ενα τετοιο λοιπόν γιατί δεν, δεν συμπεριλαμβάνει ένα κανόνα. Η επιλογή θα ήταν να υπάρχει ένας κανόνας που θα ισχύει για όλα τα κρατημέλη με το, όπως υπάρχει δηλαδή στις ε, πωλήσει online, να υπάρχει ένα, μία ε, περίοδος όπου θα ισχύει για κάθε σύμβαση. Νομίζω ότι έτσι θα ενισχύσουμε και την νομική ασφάλεια και θα επιτύχει η πρόταση και έναν από τους στόχους της. Να σταματήσει δηλαδή τον κατακαιρματισμό που υπάρχει στο συγκεκριμένο πεδίο από τα διάφορα εθνικά συστήματα. Πέμπτο και τελευταίο μου σχόλιο είναι οι ζημίες. Ε, είχα να, θα ήθελα πολλά να πω για το θέμα αυτό, αλλά η συζήτηση ήδη έγινε για κάποια σημεία, οπότε θα πω απλώς ότι συμφωνώ απολύτως με τον καθηγητή Μπίου, ότι θα, είναι αμφισβητήσιμο αν αυτός ε, ο κανόνας περιορίζει τη δυνατότητα των ε, καταναλωτών να μπορούν να αποζημιωθούν αν δεν έχει γίνει η ζημία στο ψηφιακό του περιεχόμενο, αλλά σε κάτι άλλο. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε στο γύρο των ερωτήσεων και απαντήσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Professor Και τώρα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Σμιτς από το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ, επίσης για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την ευκαιρία που μας δώσατε καλώντας μας ε, στην δημόσια ακρόαση. Εγώ δεν θα επικεντρωθώ στις προτάσεις για το ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά στις ε, προτάσεις 635 για τις συμβάσεις για την επιγραμμική πώληση αγαθών. Για το θέμα αυτό, όπως φάνηκε από τις συζητήσεις, έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες για ε, ε, για επανόρθωση, συμβατική επανόρθωση. Πρόκειται για την οδηγία 1999-44 ε, που δίνει αυτά δικαιώματα και αποτελεσματικά δικαιώματα να ζητήσουν αντικατάσταση, επισκευή, ε, μείωση τιμής ή και τερματισμό μέσω καταγγελίας της σύμβασης προϊόντων που αγοράζονται είτε επιγραμμικά είτε σε ένα κατάστημα. Η οδηγία αυτή που θεσπίστηκε πριν από 10 χρόνια οδήγησε σε πολλές ε, αλλαγές στην ε, εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έγινε μία από τι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις ε, για το ενοχικό δίκαιο. Το ίδιο και σε άλλα Θα ήθελα να τονίσω εδώ τη σημασία που έχει αυτή η πρόταση, γιατί η τωρινή πρόταση θα αναγκάσει και πάλι τα κρατημέλη να προσαρμόσουν το ενοχικό του δίκαιο σε μεγάλο βαθμό στι νέε διατάξει τη οδηγία. Τώρα, ως προς την πρόταση, θα σχολιάσω την πρόταση, τη πρόθεση, πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει τρία διαφορετικά πράγματα. Καταρχήν για τις εξαποστάσεις πωλήσεως και όχι για τις πωλήσεις με φυσική παρουσία των συμβαλωμένων, αλλά για προστασία το, της προστασίας για υπάρχοντα δικαιώματα από ελάχιστα ως πλήρη εναρμόνιση και θα δείτε ε, την πρώτη και θα παρέλθω αργότερα στη δεύτερη συνέπεια, δεύτερο στόχο τη πρόταση είναι να αλλάξει κάποιου από τους κανόνες ουσιαστικού δικαίου για, τις συμβατικές, ε, για τα συμβατικά μέτρα επανόρθωση. Θα τα βρούμε και αυτά στι στις και επίσης διευκρινήσει που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα υπάρχοντα δικαιώματα. Θα το δείτε, βλέπετε κάποια παραδείγματα στις διαφάνειες και μάλιστα τα διεξοδικά μου σχόλια θα τα βρείτε στο έγγραφο και αν το διαβάσατε θα διαπιστώσετε ότι είμαι πολύ θετικός για το τρίτο σημείο της διευκρίνησης των υφισταμένων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη, και σημαντική αυτή η διευκρίνηση γιατί στην καθημερινή πρακτική μερικά από τα σημεία που βλέπετε στις διαφάνειες ήταν ασαφή ε, από την παρούσα οδηγία για τις ε, ε, πωλήσει καταναλωτικών αγαθών. Και η νομολογία διευκρινίζει κάποια σημεία, αλλά όχι όλα. Οπότε, όση μεγαλύτερη σαφήνεια, τόσο το καλύτερο. Για τι άλλε δύο καινοτομίε τη νέα οδηγία είμαι πιο επικριτικό. Οπότε, στα 7 λεπτά που μου απέμειναν, θα ήθελα να σα αναλύσω τι βασικέ μου κριτικέ παρατηρήσει και να υποβάλω και κάποιε συστάσει προ την Επιτροπή σα. Τέσσερα σχόλια έχω συνολικά. Το πρώτο ε, είναι και το κεντρικό. Η παρούσα πρόταση θα μειώσει την περιπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι οι πολιτές θα πρέπει να μπορούν να απολούν στις, ε, στους ε, καταναλωτές με βάση τους ίδιους συμμετικούς κανόνες. Κάτι που δεν ισχύει τώρα, γιατί μια επιχείρηση που εδράζει στη χώρα Α θέλει να πωλήσει στην, ε, σε καταναλωτές στη χώρα Β θα πρέπει να λάβει νομικές συμβουλές για τις διαφορές των νομικών ε, ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά το επίπεδο προστασία του καταναλωτή. Ακριβώ για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα προτείνει εναρμόνιση όλων των μέτρων επανόρθωση των συμβατικών. Βέβαια, η παρούσα πρόταση θα συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στη μείωση τη περιπλοκότητας και του κατακαιρματισμού για συγκεκριμένα θέματα, αλλά Έχω και δύο βασικούς λόγους για αμφιβολία. Για παράδειγμα, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφήνει πολλά σημαντικά θέματα κατά μέρους που ήταν ε, στην ε, πρόταση του 2011 για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δικαίου, ε, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων, όπως ζημίες για μη εκπλήρωση της υποχρέωσης ή μη σωστή ενημέρωση για το περιεχόμενο. Και για τα θέματα αυτά θα πρέπει και πάλι να ενημερώνεται ο πολίτης για το όλο το δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλήξει σε είδους συμβατικούς όρους για τις εχώρες και τις διασυνοριακές πωλήσει δεύτερος λόγος αφιβολίας που είναι ακόμη πιο σοβαρός. Η πρόταση ε, συμβάλλει στην παρουσ... στον παρόντα κατακαιρματισμό των συμβατικών επαναρθώσεων, γιατί μιλάει μόνο για τις εξαποστάσεις πωλήσει, γιατί αφαιρεί από το πεδίο εφαρμογής ε, τις offline πωλήσει. Της οδηγία, την οδηγία δηλαδή 9944 που μέχρι τώρα ίσχυε σε όλες τις συμβάσεις καταναλωτικών αγαθών. Οπότε θα πρέπει για τις offline πωλήσει να ισχύουν άλλες διατάξεις. Οπότε δεν έχουμε ίδιες διατάξεις συμβατικές για τις εξαποστάσεις πωλήσει και τις πωλήσει που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο, με φυσική παρουσία των αντισυμβαλωμένων. Οπότε υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει κατακαιρματισμός του νομοθετικού πλαισίου βλέπετε ε, μέτρα επανόρθωσης ε, για τις ε, συμβάσει με φυσική προεσία καλύπτονται από την οδηγία για την Προσία του καταναλωτή, ενώ η νέα οδηγία καλύπτει μόνο τις επιγραμμικές πωλήσει. Ό,τι αφορά τις επανορθώσεις για τις εξ αποστάσεις πωλήσει εφαρμόζεται η οδηγία του 95 και το εθνικό δίκαιο και για το ψηφιακό περιεχόμενο ισχύει η πρόταση 635. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιες είναι οι συστάσεις μου προκειμένου να αλλάξει η παρούσα πρόταση, έχω τρεις διαφορετικές συστάσεις. Η πρώτη είναι να ε, περιληφθούν και οι στάσεις με φυσική παρουσία των αντισυμβαλωμένων ε, στην πρόταση αυτή. Να μην εκπέσουν από το πεδίο εφαρμογής και να μην περιμένουμε την ανάλυση της καταλληλότητας της πρότασης. Επίσης, να υιοθετηθεί ένα πιο λεπτομεριακός και εξεζητημένος κατάλογος ε, προϋποθέσεων περιλαμβάνοντας και τις αξιώσεις της αποζημίωσης. Και τρίτη σύσταση, ε, με δυσαρεστή που το κάνω, αλλά είμαι εδώ ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και όχι ως πολιτικός, γι' αυτό και το εντοπίζω, για να αντιμετωπιστεί η περιπλοκότητα και να διευκολυθεί η εφαρμογή στα κράτη-μέλη, διαρωτώ με μήπω θα έπρεπε να σκεφτούμε πιο αναλυτικά την επιλογή των διαφόρων ε, του, του κατάλληλου μέτρου. Θα είναι κανονισμός, θα είναι ένα προαιρετικό ε, μέσο, μήπως ε, καλύτερο στην περίπτωση αυτή. Αν διαβάσετε το εγγραφό μου λέω ότι είναι φιλόδοξες οι δύο προτάσεις. Ίσως έχει ε, νόημα να δείξουμε μια φιλοδοξία νομοθετική, αλλά όπω και στην οδηγία του 99, τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν τεράστιο κόστο για να εφαρμόσουν στην ενωμή του τάξη την οδηγία αυτή που αγγίζει την καρδιά του ιδιωτικού δικαίου. Και αναρωτιέμαι αν αξίζει τελικά τον κόπο η όλη προσπάθεια, δεδομένου του υψηλού κόστου. Σε ό,τι αφορά του κανόνε ουσιαστικού δικαίου που προσθέτει, το σημείο 2 αφορά με την ε, μετατροπή των υφισταμένων δικαιωμάτων σε ένα καθεστώς μέγιστης εναρμόνισης. Και επίσης ε, τη δυνατότητα να υπέχει ε, ευθύνη ο πολιτής για έλλειψη εκπλήρωσης και επίσης η διετής περίοδος ε, ε, μετατρέπεται σε καθεστώς μέγιστης εναρμόνιση. Τεράστια αλλαγή. Και αν λάβουμε υπόψη τα πρότυπα συμμόρφωσης, ε, θα πρέπει τα αγαθά να πληρούν τις, την κανονι, τις, τους όρους κανονικής χρήσης που αναμένει ο καταναλωτής. Και ειδικά τα μη αναλώσιμα αγαθά θα πρέπει να διαρκούν πολύ περισσότερο από μία διετία. Αν αγοράσω ένα πλυντήριο, αν αγοράζω ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο ή μια οικιακή συσκευή, Ίσως όμως αντιμετωπίσω ένα ελάττωμα που θα εμφανιστεί μετά από μια διετία. Ενώ η εύλογη προσδοκία του καταναλωτή είναι ε, η συμμόρφωση να καλύπτει μια τριετία και τετραετία. και αυτά τα θέματα για τα μη αναλώσιμα αγαθά που δεν ε, αγοράζονται επιγραμματικά, τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι καλύπτεται. Επίσης, ε, δεν είμαι υπέρ της μέγιστης εναρμόνισης στο άρθρο 14 της πρότασης. Το τρίτο σημείο, μου έμεινε ένα λεπτό, αφορά την καταγγελία της σύμβασης, τον τερματισμό. Δεν θα πω τίποτα επιπλέον για την δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης και σε περίπτωση ίσονος ελαττώματος. Θα πω κάτι άλλο. Η πρόταση δεν έχει ε, άλλο κανόνα για τις αποζημιώσεις ή πέραν της ε, καταγγελίες. Οπότε όταν έχουμε σοβαρή ε, έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός από τον τερματισμό, την καταγγελία της σύμβασης, θα πρέπει να μπορεί να δικαιωθεί και αποζημίωση. Δηλαδή, αν αποφασίσει να καταγγείλει ο καταναλωτής της σύμβασης, αλλά μόνο ε, αν μπορεί να αγοράσει αλλού και σε υψηλότερη τιμή το ίδιο προϊόν, ο πολιτής και ο καταναλωτής θα πρέπει να αναλύουν το εθνικό δίκαιο για να δει τι αποζημίωση δικαιούται σε τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη εναρμόνισης των απαιτήσεων αποζημίωσης δεν είναι πιστικά. Και η δική μου σύσταση είναι να προσθεθεί μία, ε, μία διάταξη και περί, ε, και περί σε περίπτωση καταγγελίας. Τώρα, το τελευταίο σχόλιο θα το αφήσω κατά μέρους και θα καταλήξω στο συμπέρασμα ότι φυσικά εκτιμώ ιδιαίτερος τις προτάσεις και τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρώ ότι η πρόταση, αν θέλει να ανταποκριθεί στη φιλοδοξία της απλούστευσης του ισχύου του σωμικού πλαισίου, θα πρέπει να είναι ευρύτερη και να καλύπτει περισσότερα στοιχεία. Σας ευχαριστώ κύριε Σμίτ για τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε ένα δεκάλεπτο μόνο για τη συζήτηση πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα με τους επόμενους εμπειρογνώμονες. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε το λόγο να υποβάλει ερωτήσεις. Mr. Ο κύριος Αξελβός. Θα ήθελα να επανέλθω στις συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου. Εδώ η αντιπαροχή είναι η παροχή των δεδομένων, η θέση ε, των δεδομένων στη διάθεση του παρόχου. Ποια είναι η φύση αυτής της σύμβασης. Θεωρείται σύμβαση αγοραπολισίας ή σύμβαση ανταλλαγής. Γιατί ανάλογα με το χαρακτηρισμό ίσως καταλήξουμε σε διαφορετικές ένομες συνέπειες. Γιατί άλλο αγορά, άλλο ανταλλαγή. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, ε, στο εξή πρόβλημα. Μέχρι στιγμής είχαμε μόνο ένα νόμισμα με το οποίο καταβάλαμε το τίμημα. Τώρα ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές που διατείνονται ότι τα δεδομένα είναι το νέο νόμισμα στον ψηφιακό κόσμο. Βέβαια θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να ε, πραγματοποιηθεί μετάβαση από το ένα νόμισμα στο άλλο. Αλλά ποια θα είναι η φύση των νέων συμβάσεων. Το συμβάσιο δηλαδή παροχή θέση σε διάθεση των δεδομένων, που κατά τη γνώμη μου είναι περισσότερο σύμβαση ανταλλαγή παρά σύμβαση αγοραπολισία. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους δύο εμπειρογνώμονες. Είναι πραγματικά πολύ ξεκάθαρα τα όσα μα είπανε και είναι πραγματικά πολύ καλά προετοιμασμένοι. Δεν το έχουμε συχνά αυτό, δεν μας συμβαίνει, γι' αυτό θα ήθελα να το τονίσω όλος ιδιαίτερος. δεν μπορώ να, να μιλήσω να πω στον κύριο Στάντον Μαϊάρ ότι η Ρώμη 1 είναι μια πολύ σημαντική σύμβαση για τους καταναλωτές και να την ε, καθιστούμε παροχημένη από την πίσω πόρτα νομίζω ότι δεν είναι πολύ σωστός χειρισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ανήκει στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε θα πρέπει την επιχειρηματολογία σας εκεί να την ξανασκεφτείτε ίσως. Για αυτά που ακούσαμε τώρα μόλις. Ένα ερώτημα και για τους δύο. το θέμα αυτό των δεδομένων ως ε, νόμισμα. Με, με ενοχλεί αυτό πολύ, γιατί τα δεδομένα είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό νόμισμα. Σημαίνουν την ταυτότητα των ανθρώπων. Αν αυτά τα δεδομένα τα δώσουμε σε κάποιον, του δίνουμε δύναμη πάνω μας. Γι' αυτό θα ήθελα εκεί να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά και να αποφύγουμε όλα όσα θα μπορούσαν να μας, να μας οδηγήσουν στο να θεωρήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα αποτελούν ένα είδος νομίσματος. Αυτή είναι μια αρχή που είναι απαράβατη για μένα. Γιατί τα δεδομένα, όποιος έχει τα δεδομένα των ανθρώπων έχει και τη δύναμη πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Ε, και επίσης να σας ρωτήσω το εξής, γιατί το είπατε Ένα λεπτό έχω σημειώσει τόσα πράγματα εδώ που δεν ξέρω πού ακριβώς το, το σημείωσα και πού το είπατε. Ε, για την κυρία Μακ, το ερώτημα που θέσατε και εσείς για το σημείο αυτό θα μπορούσατε ίσως να μου το διευκρινίσατε. Ευχαριστώ. Mm. Κυρία Ρέδα, σύντομο ερώτημα. Ναι, συμφωνώ με αυτά που λέει η κυρία Γκέπχαρτ για την ποιότητα των ε, παρουσιάσεων σας. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μας και για τη δουλειά που κάνουμε. Έχω ένα ερώτημα ε, ως ε, συνέχεια της παρουσίασης της κυρίας Μακ είπατε ότι είναι ασαφές αν η διάταξη για, ε, για τα δικαιώματα από τον καταναλωτή στον, θα, θα, μπορεί να λειτουργήσει ως θέμα ευθύνης αν δεν μιλούμε για προσωπικά δεδομένα. Αν κάποιος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ας πούμε τις πληροφορίες μας, βάζω εγώ ας πούμε τις, τις φωτογραφίες μου στο, στο στο ε, Facebook. Ε, μεταφέρω το δικαίωμα χρήση των, ε, φωτογραφιών μου στο Facebook. Και μετά του λέω ότι θέλω να, διαγραφούν αυτές οι, οι φωτογραφίες. Αλλά αν δεν υπάρχει θέση παναχώρησης, κανείς δεν θα μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει. Δεν δημιουργούμε ένα νομικό κενό έτσι. Δηλαδή κάποιες πληροφορίες θα είναι παντελώς μη... Ε, θα είναι εντελώ αδύνατο να χρησιμοποιηθούν. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους προσδεκλημένους μας για να απαντήσουν. Um, thank you for... Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα είμαι σύντομη. Καταρχάς, για το κατά πόσο το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να αποτελέσει ε, μέρος ε, σύμβασης που διέπει το ανταλλακτικό εμπόριο και όχι το εμπόριο πώλησης με χρηματικό αντίτιμο. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το αποφασίσει αυτό, ωστόσο όταν μιλούμε για B2C συμβάσεις, συμβάσεις επιχειρήσεων προς καταναλωτές, το θεωρώ περίεργο να θεωρηθεί ότι ένας καταναλωτής ε, προβαίνει σε ανταλλακτική συναλλαγή με μια επιχείρηση. Από εκεί και πέρα εξαρτώνται όλα αυτά και με τις προσδοκίες ε, που έχει κανείς και αυτό συνδέεται και με το ερώτημα της κυρίας Κέπχαρτ ως προς την αξία των δεδομένων. Προσωπικά πιστεύω ότι τα δεδομένα είναι εξαιρετικά σημαντικά για τους ανθρώπους, για τον κόσμο και ε, αυτός που τα συλλέγει σίγουρα έχει και ορισμένη εξουσία εναντί των ανθρώπων. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει οι προσδοκίες μας να είναι πολύ υψηλές σε σχέση με αυτά που λαμβάνουμε σε αντάλλαγμα για τα δεδομένα. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και των κανόνων ε, του εναρχικού δικαίου, για τις συμβάσεις, του δικαίου των συμβάσεων. Και τέλος για τη μεταφορά του copyright. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να αποφύγουμε νομικά κενά. Πράγματι, η οδηγία αυτή πρέπει να ξεκαθαρίσει τι είδου ανταλλαγή δεδομένων εμπίπτει ε, στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ευχαριστώ. Και ο επόμενος ε, ομιλητής, και εγώ δεν έχω πολλά να απαντήσω, το θέμα του ορισμού είναι πολύ σημαντικό και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποια είδη συμβάσεων καλύπτονται από αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ε, πρέπει να το απαντήσει αυτό. Ε, Δόκτωρ Στάντον Μάιερ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ε, σύμβασης αγοράς, η σύμβαση ανταλλαγής. Ε, αυτό που λέμε εδώ είναι ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και μπορούν να ορίσουν ε, την σύμβαση όπως οι εθνικοί τους, οι εθνικοί τους κανόνες το προβλέπουν. Δεν θέλουμε να παρέμβουν, να σε αυτό, αλλά συμφωνώ και με εσάς και με την κυρία Γκέφχαρτ για τη σημασία που έχουν τα δεδομένα. Εγώ το είπα, το εξήγησα με το νόμισμα του αύριο, αλλά τα δεδομένα σας προφανώς είναι κάτι διαφορετικό από νόμισμα. Και απαντώ έτσι και στο ερώτημα της κυρίας Ρέντα. Ε, εδώ μιλούμε για ε, πληρωμή, ε, πληρώνουμε δηλαδή με ευρώ κανονικά τα χρήματα, αλλά θα μπορούσαμε ψηφιακά να πληρώσουμε με bitcoins και μετά με δεδομένα. Τα δεδομένα δεν είναι το ίδιο με τα χρήματα, αλλά είναι μία αντιπαροχή και, τα δύο, ε, και οι δύο νομικές ας πούμε, καταστάσεις προέρχονται από δύο διαφορετικές ε, ε, περιπτώσεις. Θέλουμε να έχουμε μία παροχή και μία αντιπαροχή. Το, δικαίωμα το δίκαιο προσθέσεις δεδομένων εξακολουθεί να, να ισχύει και πρέπει γιατί προέρχεται από, το, από τον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οπότε δεν είναι θέμα να έχω εγώ εξουσία ή μη ενός τμήματος της προσωπικότητάς μου. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει για την προσθέση δεδομένων γιατί προκύπτει προφανώς από, την, ε, από τη θεμελιώδη αυτή αρχή. Τώρα, για το ε, ε, περιεχόμενο στο, στο διαδίκτυο, μιλούμε για φωτογραφίες για παράδειγμα. Αν εγώ μέσω του cloud δώσω μια φωτογραφία μου, η οποία όμως δεν μπορεί να συνδεθεί με μένα. Είναι μια φωτογραφία ενός βουνού που έβγαλα στις διακοπές μου, δεν μπορεί να τη συνδέσει κανείς με μένα. Αυτό ισχύει ως αντιπαροχή γιατί ο πάροχος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη φωτογραφία του δικού μου του βουνού για να κάνει διαφήμιση. Όλα όμως αυτά υπάρχουν και εμπίπτουν στην οδηγία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 10 λεπτά η κυρία Μπενεντίκτ Φοβάχκ Κοσούν από το Πανεπιστήμιο Πάνθεων Παρίσι 2. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο σήμερα το απόγευμα. Θα είναι πολύ σύντομη η παρουσίασή μου. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για την επανόρθωση και για την καταγγελία η λήξη της σύμβασης σε περίπτωση παροχής ψηφιακού περιεχομένου, αλλά και για την τροποποίηση της σύμβασης. Και θα ασχοληθώ μόνο με τα συγκεκριμένα κείμενα της οδηγίας. Άρθρα 13, 15 και 16. και ε, σύντομα θα δείτε την παρουσίαση στην οθόνη. Λήξη ή καταγγελία, termination, είναι ο τίτλος του άρθρου 13 και πιστεύω ότι ο όρος termination είναι παραπλανητικός γιατί η καταγγελία προβλέπεται όταν υπάρχει επανόρθωση λόγω έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση και θα πρέπει αυτό να το εξετάσουμε με το, σε αντιπαραβολή με το, 2000, με το, άρθρο, με το άρθρο 16. Επομένως, εάν ένας καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος, μπορεί να προσφύγει στο άρθρο 13, να βασιστεί σε αυτό, αλλά μπορεί επίσης να βασιστεί στο άρθρο 16, όμως μόνο εάν έχουν μεσολαβήσει, αν έχουν μεσολαβήσει 12 μήνες. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι το άρθρο 13 για την καταγγελία η λήξη της σύμβασης θα πρέπει να ερμηνεύεται από κοινού με το περιεχόμενο του άρθρου 11 με τίτλο «Επανόρθωση λόγω ε, αποτυχίας παροχής του ε, περιεχομένου. Εάν δηλαδή ο προμηθευτής δεν προμηθεύει, τότε ο καταναλωτής έχει άμεσο δικαίωμα να ε, λήξει το, τη σύμβαση, και το οποίο, ε, πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το άρθρο 13 είναι εξαιρετικά διαφορετικό, γιατί όταν ε, ο προμηθευτής δεν είναι ότι δεν προμηθεύει, αλλά προμηθεύει χωρίς να συμμορφούται η καταγγελία είναι στο τέλος Μπορεί κανείς να καταγγείλει και να λήξει τη σύμβαση μόνο εάν ο προμηθευτής τελικά δεν κατάφερε τη σύμβαση να την κάνει να συμμορφούνται με τις προδιαγραφές. Και άρα αποδυναμώνεται η προστασία του καταναλωτή στις χώρες όπου δεν υπάρχει ιεραρχία στα μέσα επανόρθωσης, όπως μας ανέφερε και ο καθηγητής κ. Χιου Μπίλ, κάτι το οποίο ισχύει και στο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Μία πρώτη παρατήρηση λοιπόν είναι αυτή και είναι πολύ σημαντική. Εάν όμως υπάρχει ιεραρχία προτεραιότητας στα μέσα επανόρθωσης, τότε η διαχωριστική γραμμή θα πρέπει να είναι ε, μεταξύ της πλήρους αποτυχίας προμήθευσης του αγαθού από τη μία και η έλλειψη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές από την άλλη. Εάν το δεύτερο εδεχόμενο είναι, ε, πλησιάζει τόσο πολύ στο πρώτο, θα μπορεί ο καταναλωτής να, καταγγείλει τη σύμβαση βάσου του άρθρου 11. Δηλαδή όταν ο, ε, προμηθευτής δεν συμμορφούται και μάλιστα η μη συμμόρφωση είναι τόσο κατάφερη, κατάφορη που να ισοδυναμεί σχεδόν με αποτυχία προμήθευσης ε, του αγαθού. Εγώ νομίζω ότι όταν έχουμε μεγάλη απουσία ε, συμμόρφωσης θα πρέπει να μην υπάρχει ιεραρχία στα μέσα επανόρθωσης, δηλαδή προτεραιότητα του ποιο θα υπερτερεί εναντί του άλλου. Και συμφωνώ με τα λεγόμενα του καθηγητή κυρίου Μπίλ. Εάν δούμε τώρα το άρθρο 13, τότε πρέπει να εξετάσουμε και το άρθρο 12 στο εδάφιο 5, το οποίο μιλά για τα μέσα επανόρθωση σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης κατά προτεραιότητα και στο 12.5 λέει ότι ο καταναλωτής δίνεται να καταγγείλει τη σύμβαση μόνο εάν η έλλειψη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της σύμβασης πλήττει τη διαλειτουργικότητα, τη λειτουργικότητα και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την παροχή της, ε, του αγαθού σε ψηφιακό περιεχόμενο. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς να προσφύγει στο άρθρο 13. Και υπάρχει και κοινοποίηση, γνωστοποίηση. Σε ορισμένες χώρες μπορεί να ισχύει αυτό. Σε άλλες χώρες μπορεί να καταγγελθεί η σύμβαση μόνο ενώπιον των δικαστηρίων. Η Γαλλία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που ε, προβλέπει ε, τη δικαστική οδό για την καταγγελία της σύμβασης. Και τώρα έχουμε μεταρρυθμίσει τον νόμο τον Οκτώβριο του 2016. Θα προβλέπεται στην γαλλική νομοθεσία η μονομερής καταγγελία και άρα λήξη της σύμβασης. Είναι δύσκολο να συμβαδίσει η καταγγελία διαγραπτής ειδοποίησης ή γνωστοποίησης και η καταγγελία της σύμβασης βάσει δικαστικής απόφασης. Και τα κράτη-μέλη θα το αποφασίσουν αυτό. Και μπορεί να αποφασίσουν τελικά τα κράτη-μέλη μόνο δικαστικά να μπορεί κανείς να καταγγείλει τη σύμβαση. Ένα άλλο ζήτημα που δεν απασχολεί την οδηγία είναι ποια είναι η προθεσμία για την κοινοποίηση ή γνωστοποίηση. Ε, και πώς θα γίνεται η ενημέρωση του εταίρου συμβαλόμενου μέρους ότι το πρώτο συμβαλόμενο μέρος καταγγέλει τη σύμβαση. Πιστεύω ότι θα δοθούν ορισμένες λεπτομέρειες ως προς το χρονοδιάγραμμα, τη χρονική προθεσμία κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί το ένα μέλος, το ένα μέρος της σύμβασης να γνωστοποιήσει στο άλλο ότι την καταγγέλει. Τώρα το δικαίωμα ε, καταγγελία η ληξεις μακροπροθεσμων συμβασεων εδω ειναι κάπω παραπλανητικη η διαταξη στο άρθρο 16. Προφανώ όταν υπογραφεί κανεί μια σύμβαση έχει το δικαίωμα να, τη λήξει. Δεν είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο δικαίωμα. Δεν μπορεί κανεί να καταδικαστεί υποχρεωτικά να παραμείνει ατέρμονα και ατελείωτα στην οποιαδήποτε σύμβαση. Λέει όμω το κείμενο ότι ο καταναλωτή δεν δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν περάσουν 12 μήνε και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε σε όσους ανησυχούν για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Εάν είναι πλήρως απούσα η συμμόρφωση, γιατί να μην μπορεί ο καταναλωτής να καταγγείλει τη σύμβαση πριν την, το πέρας των 12 μηνών. Αυτό ισχύει διότι ε, όταν κανείς υπογράφει μία σύμβαση, ενδεχομένως στην αρχή της, ε, λαμβάνει κάποια αγαθά, π.χ. ένα τηλέφωνο θα, πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ε, εκεί. Υπάρχουν άλλες συμβάσεις που δεν λαμβάνει τίποτα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λογικό να μην μπορεί κανείς να καταγγείλει μια σύμβαση πριν το πέρας 12 μηνών, μόνο αν έχει λάβει αγαθά στην αρχή της σύμβασης, π.χ. ένα τηλέφωνο. Εάν μπαίνει σε μια σύμβαση, δεν, δεν, δεν λαμβάνει τίποτα στην αρχή και υπάρχει πλήρης απουσία συμμόρφωσης, δεν ε, ε, λαμβάνει το αγαθό της σύμβασης, γιατί δεν μπορεί να την καταγγείλει από την αρχή. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των δύο. Και δεν μπορώ, είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να πούμε ότι οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις είναι αυτές που ξεπερνούν τους 12 μήνες. Και αυτό είναι απαραίτητο για τη διευκρίνηση. Τέλος, να σας πω δύο λόγια για το άρθρο 15, το οποίο είναι αφορά στην τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου. Μιλούμε για την τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου από τον πάροχο της υπηρεσίας ή το προμηθευτή του αγαθού, όχι από τον καταναλωτή. Δηλαδή μόνο ο πάροχος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιφερειεχόμενο, κάτι το οποίο είναι κατανοητό γιατί εξελίξει εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Ωστόσο, οφείλουμε να αναρωτηθούμε το άρθρο 15 πόση εξουσία δίνει στον κλάδο στη βιομηχανία. Μήπως δίνει υπερβολικά πολλή εξουσία και θα μπορεί μετά η βιομηχανία αυτή μονομερός να τροποποιήσει τη σύμβαση. Και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο το άρθρο 15 θα ισχύει εάν ο καταναλωτής έχει την επιλογή της αναβάθμισης και αυτό ίσως είναι επικίνδυνο για ορισμένους καταναλωτές. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά σαφή. Τέλος, ε, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ε, θεωρώ ότι αυτές είναι πολύ σημαντικές διατάξεις και δυσνόητες στην πρώτη ανάγνωση της οδηγίας. Ίσως γιατί δεν έχει γίνει αρκετή ε, δουλειά έτσι ώστε στους τίτλους ε, για να φανεί η διαφορά μεταξύ του άρθρου 11, του άρθρου 13 και του άρθρου 16. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα δεκάλεπτο τώρα για περαιτέρω συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο παρόντες ευρωβουλευτές, αλλά και βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων. Και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η κυρία Πάκο από την BUC, η κυρία Μάινς από την Αυστρία, από το εμπορικό επιμελητήριο της Αυστρίας, μήπως θα ήθελαν να λάβουν το, το λόγο, η κυρία Πάκο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που δίνεται στις ε, ενώσεις καταναλωτών να συμβάλλουν στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση που γίνεται στην απογευματινή δημόσια κρόση, το εργαστήριο. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα αναφέρθηκα, δεν ξέρω πώς χρόνο έχω. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική και να επικεντρωθώ στις βασικές μας ανησυχίες και στο βασικό μας προβληματισμό. Εν συντομία λοιπόν, καταρχήν χαιρετίζουμε τη μετάβαση από την προαιρετική εναρμόνιση που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινό Δίκαιο Πολίσεων στην πιο στοχευμένη εναρμόνιση μέσω οδηγιών που έχει πιο υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δεν έχουμε πρόβλημα με τη μετάβαση αυτή. Πρόβλημα έχουμε όμως με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει πλήρη εναρμόνιση αποκλείοντας εθνικές νομοθετικές διατάξεις που έχουν άλλο επίπεδο εναρμόνισης ε, ή αποκλεί τέτοια δυνατότητα στο μέλλον. Κάτι που σημαίνει ότι σε μερικές ε, χώρες μέλη οι καταναλωτές στερούνται εξαιτίας αυτής της τελευταίας πρότασης κάποια δικαιώματα που είχαν στο παρελθόν από την Εθνική ε, Νομοθεσία και δεν πρόκειται για ασήματα δικαιώματα αλλά για ε, βασικά δικαιώματα μακράς νομικής παράδοσης και κάτι τέτοιο ενοχλεί ιδιαίτερως τους καταναλωτές και τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν. Επίσης θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβαλε τον αντίκτυπο του κανονισμού Ρώμη 1, ιδιαίτερα το καθεστώ των καταναλωτών, λέγοντα ότι οι πολιτέ είναι υποχρεωμένοι να μελετούν το, νομικό, το εθνικό δίκαιο και να προσαρμόζουν του συμβατικού όρου πριν επεκτείνουν τις πωλήσει του σε άλλα κρατημέλη. Δεν ισχύει αυτό, ούτε από νομική, ούτε και από πρακτική άποψη, γιατί ο κανονισμός Ρώμη 1 επιλέγει, ε, επιτρέπει την επιλογή δικαίου ακόμη και για τις ε, συμβατικέ ενοχές. Και αυτό κάνουν οι πολίτε και συνήθω επιλέγουν το κράτος, το, δίκαιο της χώρας τους. Και αυτό, αυτή η δυνατότητα επιλογής ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Και όπως είπαν και πολλοί εμπειρογνώμονες, ίσως δεν θα έχουμε με αυτόν τον τρόπο την αναμενόμενη αύξηση των διασυνοριακών ε, δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να έχουμε μια αναλογία και εξισορρόπηση των θυσιών που θα κάνουν οι καταναλωτές σε ορισμένες χώρες ε, με τα κέρδη και τα συμφέροντα των πολιτών. Ε, ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Στάντερ Μάιρ, ε, με προβλημάτισε κάπω, γιατί είπε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον μόνο το 1% των καταναλωτών επηρεάζονται. Ξέρουμε ότι μετά από 6 χρόνια ή μέσα... για 6 χρόνια μπορούν να, να επισημάνουν ελαττώματα στο αγαθό που αγόρασα και να ζητήσουν αποζημίωση. Δεν νομίζω ε, ότι η προσέγγιση όταν ο καταναλωτής δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του είναι σαν να μην τα έχει. Αυτό είναι λάθος. Για παράδειγμα, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού ε, οι καταναλωτέ ασκούν τα δικαιώματά του. 51% των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα σε ό,τι αφορά τις πωλήσει ε, προϊόντων και πιστεύουν ότι η συμμόρφωση θα πρέπει να ισχύει ε, όσο εύλογα περιμένει κάτι τέτοιο καταναλωτή. Όταν αγοράζει κανεί ένα πλυντήριο δεν περιμένει μέσα σε δύο χρόνια να χαλάσει. Θα πρέπει να ισχύει η δυνατότητα ε, και το δικαίωμα αποζημίωση και μετά τη διετία. Για παράδειγμα, ο, ο διαμεσολαβητής, ο συνήγορος του πολίτη, έχει λάβει πολλές ε, αιτιάσεις, πολλά παράπονα από καταναλωτές που αγόρασαν ε, προϊόντα και τα ελαττώματα φάνηκαν μετά, μετά τη διετία. όλοι αυτοί θα χάσουν τέτοια δικαιώματα στο μέλλον, γιατί δεν θα ισχύει μεγαλύτερη προθεσμία. Επίσης, η διάκριση μεταξύ επιγραμμικών και offline πωλήσεων θα μπερδέψει τους καταναλωτές, γιατί ισχύουν διαφορετικά δικαιώματα σε διαφορετικές χώρες για τα offline και τα online. Και 80% των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο είπαν ότι στο μέλλον θα αγοράζουν μόνο από καταστήματα. Δεν πρόκειται να αγοράζουν ε, στο διαδίκτυο αν τα δικαιώματά τους εξασφαλίζονται καλύτερα από πωλήσει στα καταστήματα. Κάτι που δείχνει κάποιες πρακτικές πτυχές ε, των αντιλήψεων των καταναλωτών και το τι θα συμβεί σε περίπτωση που ε, υποβληθεί αμετάβλητη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Μάινς, μήπως εσείς θα είχατε καλοσύνη να είστε πιο λακωνικοί, γιατί στο μεταξύ και δύο άλλοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο και ένα πεντάλεπτο έχουμε συνολικά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Γενικώ για το δίκαιο προστασία των καταναλωτών, προ το παρόν η κατάσταση έχει ω εξή. Το δίκαιο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο από κοινού με το εθνικό δίκαιο θεωρείται ε, αρκετά περιπεπλεγμένο ε, και από τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε πάρα πολλές διασυνδεδεμένες ε, οδηγίες κανονισμούς και οι εταιρείε βεβαίως είναι ιδιαίτερως φορτωμένες με την εφαρμογή όλων αυτών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν ε, και προσαρμογές ε, και ο στόχος αυτής της ε, οδηγίας είναι να εμποδίσει ουσιαστικά να βάλει τρικλοποδιά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να θα αρχίσει να λειτουργεί το μέτρο αυτό. Έχει το στόχο να βάλει ακριβώς τρικλοποδιά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. εμπόριο. Και Έχουμε και την οδηγία για τα καταναλωτικά αγαθά, η οποία είναι ε, ε, λίγο πολύ εναρμονισμένη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη δική μας άποψη είναι απαραίτητο, επίγον ακριβώ και λόγω της περιπλοκότητας που υπάρχει του υπάρχοντος δικαίου, να, αντί να γίνει μια νέα πρωτοβουλία νομοθετικής πρότασης, να γίνει μια εις αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας. για το επίπεδο της προστασίας του καταναλωτού. Ακούω συνέχεια ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές, ε, το επίπεδο ε, δεν μπορεί να ε, μειωθεί της προστασίας. Πρέπει να πω ότι έχω μιλήσει με πολλούς εκπροσώπους επιχειρήσεων και για τα δικαιώματα των καταναλωτών και για τα αποτελέσματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή και για τις ε, πωλήσει ε, εξ και για τις ε, πωλήσει στα καταστήματα. Και πρέπει να πω ότι οι επιχειρήσεις είναι όλο και περισσότερο της άποψης ότι οι κανόνες που δημιουργούνται το τελευταίο καιρό είναι μη φιλικοί προς τις επιχειρήσεις και επίσης είναι άδικοι. Υπάρχει ανισορροπία σε πολλούς τομείς και υπάρχει, ε, αντιμετωπίζουμε ένα, μια δίνη προς τα πάνω τώρα ε, και φοβούνται οι επιχειρήσεις ότι, και λογικό ότι πέραν της ε, σημαντικής επιδείνωσης για το εις των, των επιχειρήσεων πολλαπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται ε, το άκθος ό,τι αφορά την ε, σύναψη αυτών των ε, συμβάσεων για, μέσω αυτής της συνολικής γενικής εναρμόνισης. Γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Σε αυτό φοβούνται ότι θα καταλήξει η νομοθεσία αυτή αν εφαρμοστεί οι επιχειρήσεις. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι όσο πιο αυστηρές είναι οι διατάξεις, οι νομικές διατάξεις, τόσο λιγότερες δυνατότητες έχουν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν από μόνες τους σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Δεν μπορούν να καλύψουν λοιπόν το κενό αυτό και γι' αυτό ε, θα πρέπει να υπάρξει ελευθερία προς τις επιχειρήσεις που υπάρχει και στην, θεμελιώδη χάρτα, στην χάρτα των θεμελιώδων ε, δικαιωμάτων. Να αφήσουμε δηλαδή στις επιχειρήσεις ένα περιθώριο ελιγμών, ένα περιθώριο δραστηριοποίησης. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα. Ο κύριος Λεμπρετόν έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις πολύ σύντομες στην καθηγήτρια κυρία Φοβάχκα Κοσού. Να σας πω όμως ότι ε, κάθε φορά που καλούμε Γάλλους μιλούν αγγλικά. Ελπίζω να μην τους δίνουν τέτοιες εντολές ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα γαλλικά είναι πολύ ωραία γλώσσα. Έχω μάθει ότι αντυχεί και στην Ουάσιγκτον θα μου άρεσε να αντυχήσει και να ακουστεί και στις Βρυξέλλες. Τώρα, επί της ουσίας, επικρίνεται τη διάρθρωση μεταξύ του άρθρου 11 και του άρθρου 13. πουσία συμμόρφωσης στις προϋποθέσεις και απουσία παροχής του αγαθού ή του περιεχομένου. Τι προτείνετε να διορθωθούν, να συγχωνευτούν σε ένα άρθρο. Αυτό δεν μας διευκρινίσατε. Και δεύτερη ερώτηση για το άρθρο 15. Καλώς εκτιμήσατε ότι είναι ένα άρθρο που δίνει υπερβολικά πολλά δικαιώματα στους παρόχους, στους προμηθευτές, να τροποποιήσουν μονομερώς το περιεχόμενο της σύμβασης. Δεν είναι αυτό αντίθετο με ε, το βασικό άρθρο του Γαλλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που λέει ότι η σύμβαση είναι ε, το κείμενο που διέπει τα δικαιώματα των μερών. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής από τη Βουλή των Λόρδων. Ε, σε σχέση με την μη συμμόρφωση ε, της παροχής γιατί στην περίπτωση της επανόρθωσης δεν μπορεί να υπάρξει σαφές όριο σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να έχουν οι καταναλωτές τη νομική βεβαιότητα ότι δεν θα παγιδευτούν σε αυτόν τον κύκλο αποτυχιών. Επίσης και δεύτερον γιατί να μην υπάρχει ιεραρχία ε, στα νομικά μέσα επανόρθωσης. Σύντομες απαντήσεις. Καταρχήν να σας ε, καθησυχάσω. Το Κοινοβούλιο με διαβεβαίωσε ότι μπορούσα να μιλήσω και στα γαλλικά, αλλά δεν προλάβαινα να συντάξω το κείμενο παρά μόνο στα αγγλικά και μια και τα τεχνικά κείμενα τα έχουμε στα αγγλικά ήταν πιο εύκολο για μένα και θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο και εγώ να εκφράσω και να γίνω αντιληπτή στα αγγλικά γιατί μερικές φορές οι μεταφράσεις ε, σε τέτοια τεχνικά θέματα δεν είναι και πολύ εύκολες. Θα σας απαντήσω πάντως στα γαλλικά. Ούτως ή άλλως ε, μου είναι πιο εύκολο. Ε, για τη σχέση των άρθρων 11 και 13. Με καταλάβατε θαυμάσια. Μία αναδιατύπωση το διάρθρο θα ήταν ασκόπιμη, προκειμένου να επαναφέρουμε στο σημείο 11 τις περιπτώσεις ε, ε, ε, έλλειψης ή μη συμμόρφωσης για τις πιο σοβαρές κατάφορες περιστάσεις έλλειψης ή μη συμμόρφωσης καταργώντας την ιεραρχία, όπως είπε ο καθηγητής Μπίλα. Αν καταργήσουμε αυτή την ιεραρχία που θεσπίζει το άρθρο 12, τότε δεν χρειαζόμαστε πια το άρθρο 11. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης, τερματισμού της σύμβασης είναι άμεση άσχετα με το είδος της μη εκπλήρωσης. Αν πρόκειται για απόλυτη ε, μη προμήθεια ή για ελαττωματικό προϊόν είναι το ίδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κοινό δίκαιο, το κοινό ενοχικό δίκαιο δεν συνάδει με τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές ε, του ενωσιακού δικαίου. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλύτερα αυτό το θέμα. Και διαρωτόμαστε αν έχει νόημα αυτή η ιεράρχηση των μέτρων επανόρθωσης σε περίπτωση ε, έλλειψης συμμόρφωσης. Ή αν κρατήσουμε την ιεραρχία τουλάχιστον να την περιορίσουμε. Γιατί αλλιώ θα εμπλακούμε σε ατέρμονες συζητήσεις για το αν πρόκειται για έλλειψη συμμόρφωσης ή για ε, αποτυχία συμμόρφωσης. Με ατέρμονες δίκες επίσης. Επίσης, γιατί να μην δώσουμε δικαίωμα άμεσης καταγγελίας ή άμεσου τερματισμού της σύμβασης. Γιατί να μην δώσουμε αυτό το δικαίωμα στον καταναλωτή. Δεν είναι ότι έκανε τόσα έξοδα ο κλάδος. Από τη στιγμή που υπάρχει το προϊόν, δεν είναι δαπανηρή η παράδοσή του, οπότε να δώσω αυτό το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας στον καταναλωτή. Γι' αυτό και είμαι ιδιαίτερα επικριτική για το άρθρο 16. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το άρθρο 15, ναι, η σύμβαση είναι το δίκαιο των συμβαλωμένων. Αυτό προβλέπει το γαλλικό δίκαιο και αυτό φάνηκε και ε, στο διάταγμα της προηγούμενης εβδομάδας που θα τροποποιήσει το ενοχικό δίκαιο, το συγκεκριμένο τμήμα του αστικού δικαίου. Εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίσταση με ραγδαίες εξελίξεις ε, και αυτό και χρειάζεται επικαιροποίηση. Αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και νομίζω ότι λήφθη υπόψη στο άρθρο 15. Ο μόνος φόβος μου είναι ότι πίσω αυτήν την ε, ε, ουδέτερη διατύπωση, τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου, μήπως κρύβεται κάτι υποπτό. Γιατί είναι ένα δικαίωμα που αποδίδεται μονομερός στον προμηθευτή. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει μια σωστή πλαισίωση των όρων υπό τους οποίους ασκείται το δικαίωμα. Τώρα, αυτό δεν θα το αναφέρω περαιτέρω για το άρθρο 15. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να βάλουμε περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του Λόρδου αυτό με προβληματίζει ακόμη περισσότερο γιατί πολύ φοβούμαι ότι ξέχασα την ερώτηση. Ε, θα μπορούσατε ίσως να επαναλάβετε την ερώτηση. Το τελευταίο ερώτημα ήταν το εξής. Γιατί να μην θέσουμε σαφές όριο στον αριθμό των αντικαταστάσεων ή επαναρθώσεων τις οποίες έχουν δικαίωμα οι καταναλωτές για να αυξήσουμε τη νομική τους ασφάλεια. Είναι ερώτηση για την Επιτροπή πιστεύω, λέει η κυρία ε, Κωσό. Απαντήστε σε 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε όριο Όμως είναι ένα όριο που προσαρμόζεται στα διαφορετικά προϊόντα γιατί ο χρόνος που χρειάζεται για να αποκατασταθεί η βλάβη του προϊόντος εξαρτάται από τη φύση του προϊόντος. Μιλούμε για υπολογιστή, για τηλεόραση, γιατί μιλούμε. Εύλογο χρονικό διάστημα δηλαδή, ε, το παίρνουμε αυτό από το common law και στην αιτιολογική σκέψη λέμε ξεκάθαρο ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να υπόκεινται σε επανειλημμένες προσπάθειες επανόρθωσης ή αποκατάστασης. Άπαξ και περάσει προθεσμία μπορούν πράγματι να καταγγείλουν τη σύμβαση και να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα γιατί δεν ε, διαλέξαμε μια επιλογή μέσων επανόρθωσης να έχει ο καταναλωτής και γιατί να έχουμε ιεραρχία γιατί 20 κράτη-μέλη έχουν, το έχουν εφαρμόσει αυτό από την οδηγία για τις πωλήσει. Είναι αυτό αλλά έχει αποδείξει και την αξία του στην πράξη. Και οι μελέτες για τα, για τα δεδομένα των καταναλωτών 77% δείχνουν ότι 77% των καταναλωτών θεωρούν ότι είναι λογικό ο προμηθευτής να προσφέρει αποκατάσταση, επανόρθωση, αντικατάσταση του προϊόντος πρώτα και μετά επιστροφή χρημάτων. Γι' αυτό επιλέξαμε την ιεραρχία ε, των μέσων επανόρθωσης. Ευχαριστούμε τώρα η καθηγήτρια κυρία Κριστιάνα Βέντερχοστ από το Ευρωπαϊκό Νομικό Ινστιτούτο της Βιέννης. Παρακαλούμε να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά αν αυτό είναι εφικτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που με προσκαλέσατε για να κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση της κρόση αυτής του εργαστηρίου αυτού και να συνοψίσω τα βασικά σημεία της συζήτησης. Έχουμε δύο προτάσεις οδηγίες που κατέθεσε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του, της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων που είχε αποσύρει ε, στα τέλη του 2014. Οι στόχοι όμως παραμένουν οι Αυτό που επιδιώκουμε είναι η ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου, ε, η διαμόρφωση ενός ε, περιβάλλοντος φιλικού για τις επιχειρήσεις και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτού. Θέλουμε κανόνες που να είναι φιλικοί προς τους χρήστες, να είναι ουδέτεροι από τεχνολογική άποψη και να αντέχουν στο μέλλον, να έχουν μια διαχρονικότητα. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι στόχοι είναι κοινοί σε όλους ε, ο, τους ομιλητές, όλους τους καλεσμένους, ε, υπήρχε ομοφωνία ως προς τους στόχους αυτούς. Επίσης, ε, αν κατάλαβα καλά, η κρατούσα γνώμη των εμπειρογνωμόνων ήταν γενικώ θετική ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγκατέλειψε το ενοχικό δίκαιο, αλλά κάνει μια νέα αρχή. Επίσης δίνει έμφαση στο, στο ψηφιακό σκέλος, προκειμένου να δώσει σάρκα και οστά στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Βέβαια πρόκειται για μια ενεξελίξη νομοθετική διαδικασία και ως νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση της πρότασης και για διόρθωση των αδυναμιών και των κενών της. Όλοι οι εμπειρογνώμονες που έλαβαν το λόγο στη συζήτηση εστιάστηκα στις προβληματικές πτυχές της πρότασης και στην ανάγκη διόρθωσης κάποιων ελλείψεων. Ένα ζήτημα που ανέκυψε ε, επανειλημμένο σχεδόν από όλους τους εμπειρογνώμονες ε, και σχεδόν όλους όσοι έλαβαν το λόγο ήταν η συνέπειες μιας πλήρους στοχευμένης εναρμόνισης. Δηλαδή, ε, πλήρους εναρμόνισης επιλεγμένων, ε, λίγων και συγκεκριμένων επιλεγμένων θεμάτων. Σε σχέση με την πρόταση για το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων, η νέα πρόταση έχει κάποιες ε, αδυναμίες για όλους, και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Βέβαια, η πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων επικεντρώθηκε στα θέματα των καταναλωτών ε, πυρογνώμονε εξέφρασαν την ανησυχία ότι οι κράτη-μέλη που έχουν υψηλότερο επίπεδο προστασία του καταναλωτή θα χρειαστεί με τις νέες προτάσει να περιορίσουν αυτό το επίπεδο προστασία του καταναλωτού. Ε, ιδιαίτερα αναφέρθηκε το ευρύ δικαίωμα που δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο για την ε, καταγγελία και την απόρριψη. Επίσης αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 11 χώρες σε ένα ή περισσότερα θέματα έχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Και παρόλα αυτά όμως η γενική αξιολόγηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι γενικώ το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή αυξάνεται, ενισχύεται με τις νέες προτάσεις. Βέβαια, οι εκπρόσωποι των επιχειρηματήσεων έθεσαν διαφορετική γνώμη και εξέφρασαν τις ανησυχίες ότι αυτό το αυξημένο επίπεδο προστασίας του καταναλωτού θα αυξήσει και τη γραφειοκρατία και το γραφειοκρατικό άχθος για τις επιχειρήσεις, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο καθηγητής Σμιτ εξέφρασε τις ανησυχίες ότι αυτή η πλήρη στοχευμένη εναρμόνιση ίσως δεν βοηθήσει και πολύ τις επιχειρήσεις, γιατί πολλά θέματα που είναι προσκόμματα στο διασυνοριακό εμπόριο, Δυστυχώ έμειναν εκτό του πεδίου εφαρμογή τη Νέα οδηγία. και ζήτησε ένα πιο περιεκτικό καθεστώ ε, και μάλιστα θα προτιμούσε ε, ε, ή ένα προαιρετικό μέσο ή ένα κανονισμό. Επίσης, ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε παρελειμμένως είναι ο κατακαιρματισμός το ενοχικού δικαίου για θέματα καταναλωτή. Ίσως επιταθεί αυτός ο κατακαιρματισμός, ίσως δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ της προμήθειας υλικών αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου ή να δημιουργήσει άλλο χάσμα μεταξύ ε, επιγραμμικών πωλήσεων και πωλήσεων με φυσική παρουσία των αντισυμβαλωμένων. Ίσως το δεύτερο, η εξαίρεση δηλαδή των ε, face-to-face -face πωλήσεων ε, δεν δικαιολογείται και πολλοί το δευτερο η εξαιρεση δηλαδη των face to face πωλησεων δεν δικαιολογειται και πολλοι το επισημαναν ο Δ. Στόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έπεισε ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα και όταν συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ε, μια πρόταση και ένα καθεστώς που θα συμπεριλαμβάνει και τις πωλήσει που γίνονται με φυσική παρουσία των αντισυμβαλωμένων. Σε ό,τι αφορά ε, τους ε, προτινόμενους κανόνες, πολλοί εμπειρογνώμονες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα κριτήρια ε, του καθορισμού, της συμμόρφωσης με τους όρους ε, της σύμβασης. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο, αυτή επικεντρώνεται κυρίως ε, στους όρους που παρέχει ο προμηθευτής. Και μόνο σε περίπτωση που είναι σαφή αυτή η όρη και η ε, λαμβάνεται υπόψη οι εύλογη προσδοκία, οι εύλογες προσδοκίες του καταναλωτού. Έτσι, ουσιαστικά αφήνουμε στην ψηφιακή βιομηχανία να καθορίσει τη συμμόρφωση και δεν ελέγχεται επαρκώς ε, ε, το περιεχόμενο των συμβάσεων σε περίπτωση που υπάρχουν πιθανότητες να είναι αθέμητες. Επίσης, ε, δεν δικαιολογείται υποβάθμιση της ποιότητας σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Τώρα, για την αποζημίωση. Ιδιαίτερα για την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο. Φαίνεται ότι περιορίζει τη δυνατότητα αυτή τουλάχιστον αυτό προσφέρει ε, αποζημίωση ε, για την υποβάθμιση του ψηφιακού περιβάλλοντος. Και αυτό, στο πλαίσιο της συζήτησης για την πλήρη εναρμόνιση, ίσως σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα επιδικάζουν ε, αποζημιώσεις για περιπτώσεις που κάει και το σπίτι του καταναλωτή που έχασε τη ζωή του σε ατύχημα. Ελπίζω Μα έπεισε όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το ζητούμενο ή ο σκοπό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ότι τα κράτη-μέλη θα είναι ελεύθερα από αυτή την άποψη, θα έχουν διακριτική ευχέρεια. Θα πρέπει όμω να διευκρινιστεί η διατύπωση για να αποφεύγονται παρερμηνίε. Επίση, τονίστηκε ότι οι όροι για τι προθεσμίε ίσω πρέπει να συζητηθούν πιο διεξοδικά Έχουμε από τη μια την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μην υπάρχει καμία προθεσμία για το ψηφιακό περιεχόμενο και από την άλλη πλευρά αφήνουμε ε, την ε, προθεσμία της παραγραφής στην απόλυτη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Αυτό που ίσως ήταν πιο σημαντικό είναι η διετής προθεσμία για την πρόταση για τις πωλήσει που ε, θα δημιουργήσει Διαφορέ σε σχέση με αυτό που ισχύει τώρα στα κράτη-μέλη και ίσως δημιουργήσει προβλήματα στους καταναλωτές, ιδιαίτερα για τα μη αναλώσιμα αγαθά, όπου τα ελαττώματα μπορεί να εμφανιστούν μετά από πολλά χρόνια. Πολλά σχόλια αναφέρθηκαν σε σχέση με τους κανόνες για την καταγγελία της σύμβασης, τον τερματισμό. Ίσως σκόπιμο θα ήταν να χρησιμοποιηθεί διαφορετική ορολογία για την καταγγελία λόγω ε, έλλειψης συμμόρφωσης ή για την καταγγελία σε ό,τι αφορά τη, τις μακροχρόνιες συμβάσεις. Σε ό,τι αφορά την καταγγελία λόγω θέτησης υποχρέωσης, υπάρχει το άρθρο 11 για την έλλειψη εκπλήρωσης ή για τη μη συμμόρφωση με το ψηφιακό περιεχόμενο. Οι διαφορές όμως ίσως οδηγήσουν σε μη συνεπή αποτελέσματα, σε περίπτωση ιδιαίτερα κατάφορης μη ε, συμμόρφωσης. Σε ό,τι αφορά τον κανόνα των 12 μηνών, ίσως και αυτό είχε αρνητικέ συνέπειες για τους καταναλωτές. Και το άρθρο 15 για την τροποποίηση ίσως δίνει υπερβολικές εξουσίες ε, στη, στον ψηφιακό καλάδο να τροποποιήσει μόνο μερός τους συμβατικούς όρους δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον πολύ σημαντικό γεγονός ότι μια σειρά σημαντικών θεμάτων όπως ε, το δυνητικό δικαίωμα του καταναλωτή να επαναπολύσει ψηφιακό περιεχόμενο, να κάνει ε, ε, παραπάνω από ένα download και να λάβει σημαντικές επικαιροποίησεις δεν, δεν συμπεριλήφθηκαν, αλλά επαφέθηκαν στην ψηφιακή βιομηχανία και στα δικαστήρια η καθηγητής ΜΑΚ επέσει την προσοχή μας στο γεγονός ότι η απόσυρση της συνένεσης σε ό,τι αφορά τη χρήση δεδομένων προσωπικών και άλλων και η συνάφεια τους με τους ε, συμβατικούς όρους ίσως δεν έχουν διαθετηθεί πλήρως. Οπότε η σημαντική επικάλυψη που υπάρχει μεταξύ του συμβατικού δικαίου αφενός και του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας για τα δεδομένα αφετέρου και όλες αυτές οι σχέσεις μεταξύ τους θα πρέπει να διευκρινιστούν. Πολλοί πυρογνώμονες ασχολήθηκαν με το θεμελιώδη ζήτημα του κατά πόσο η πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλη με το σκοπό που εξυπηρετεί υπό το φως και του γεγονότος ότι το περισσότερα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου δεν αφορούν μόνο δύο μέρη. Γιατί μπορεί ένας καταναλωτής να αγοράσει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ε, σε ένα κατάστημα και όταν το φορτώνει στο, με το λογισμικό στο κομπιούτερ θέλει του ζητάτε η άδεια για τον του τελικού χρήστη. Επίσης, τα περισσότερα ψηφιακά προϊόντα είναι υβριδικής μορφής σήμερα. Δηλαδή, απαιτούν συνεχή πρόσβαση σε υποδομές που συνήθως ε, είναι υποδομές ε, νεφοϋπολογιστικής. Οπότε έχουμε πολλά αντισυμβαλόμενα μέρη και πολλαπλές ε, συμβάσεις. Και εδώ είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια είναι η σύμβαση της προμήθειας και πώς ε, ε, γίνεται αντιληπτή η συμμόρφωση με τη σύμβαση και με ποια σύμβαση όταν μιλούμε για πολλαπλές συμβάσεις. Επίσης, ε, πολλοί ομιλητές μίλησαν για μία φράση που έγινε πολύ της μόδας, το διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε θα το αντιμετωπίσει σε μεταγενέστερο στάδιο αυτό το θέμα του ίντερνετ των πραγμάτων, του διαδικτύου των πραγμάτων. Βέβαια κάποια πράγματα που σχετίζονται με αυτό το, αυτή την έννοια έχουν τόσο στενή αλληλεπίδραση με την συμμόρφωση και τα μέτρα επανόρθωσης για τη μη συμμόρφωση που ίσως δεν είναι σκόπιμη αναβολή της συζήτησης για μεταγενέστερο στάδιο. Ήδη ή τώρα ή στο πολύ εγγύς μέλλον η τωρα η στο πολυ εγγυς η πλειοψηφια των αγαθών που αγοράζουμε θα έχουν ενσωματωμένο λογισμικό και ε, διασυνδεσιμότητα με το διαδίκτυο. Αυτό ήδη ισχύει με τα περισσότερα νέα οχήματα ή τσικιακές συσκευέ. Και μάλιστα το φαινόμενο αυτό θα γενικευθεί σε πολύ περισσότερες συσκευές, ακόμη και σε εξοπλισμό, σε τρόφιμα ή μέσα ένδυσης. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις θα αντέξουν το πέρασμα του χρόνου και δεν θα χρειαστούν επικαιροποίηση, δεν θα ξεπεραστούν μέσα σε μια 15 Αυτό είναι αν μη τι άλλο συζητήσιμο ε, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων. Ο χρόνος πιέζει, ελπίζω να κατάφερα να κάνω μια ανακεφαλαίωση των ε, βασικών σημείων της απογευματινής συζήτησης. Ζητώ συγγνώμη αν παρέλειψε ορισμένα θέματα. Ε, επειδή με προσκαλέσατε ως εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου που ασχολείται με το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια ε, υπό την προεδρία του Λόρτ Τόμας, ε, δικαστή ε, της Αγγλίας και Ουαλίας. Ε, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Ευελπιστώ ότι η νομοθετική διαδικασία θα καταλήξει σε χρήσιμο αποτέλεσμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους καταναλωτές, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η ψηφιακή αγορά και να δημιουργηθεί μια κατάσταση εποφελής για όλους, όπως ε, υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική της παρουσίαση. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνω αυτήν την ανακεφαλώση και ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την ε, καθηγήτρια Φάντροχόστ που συνόψισε τις, ε, τα όσα ακούστηκαν σήμερα στο εργαστήριο. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, προσκεκλημένους μας που ήταν σήμερα παρόντες, που μοιράστηκαν τις απόψεις τους μαζί μας. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή αρχή της συζήτησης για τούτες τις δύο προτάσεις οδηγιών. Να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων φορέων που ήταν σήμερα παρόντες. Ευχαριστώ βεβαίως και τα μέλη της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και τα μέλη της Επιτροπής Γιούρι. Ξέρω ότι αυτό το θέμα είναι πραγματικά ατελείωτο και ε, σίγουρα θα ξαναβρεθούμε στο μέλλον. Εγώ τουλάχιστον από την ομάδα φεύγω με περισσότερα ερωτηματικά από ό,τι ήρθα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάντα καλό. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ.